Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να ξεκινήσουμε με το σημείο 17 απευθεία στην ημερήσια διάταξη. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν την ακρόαση, στην οποία πιστεύω αποδίδουν μεγάλη σημασία τα μέλη τη Επιτροπή μα. Πρόκειται για την ακρόαση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά κάποιο τρόπο αποτελεί και την εισαγωγή στην συζήτηση για το μέλλον του εν λόγω ταμείου. Με ανάλυση του ρόλου και του, της αποτελεσματικότητας των αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των διαφόρων πρωτοβουλειών που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ τους τρεις προσκεκλημένους που ήρθαν. Θα τους δώσω αμέσως το λόγο. Προηγουμένως όμως, θα ήθελα να υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε ορίσει αφού η, η ακρόαση οργανώνεται σε δύο τμήματα, η σημερινή καταρχάς με τους ειδικού όπως τους ονομάζουμε, που θα συμπληρώσει μια δεύτερη ακρόαση, ένα δεύτερο τμήμα μάλλον ακρόαση στο Φεβρουάριο του 2011 με τους κοινωνικούς εταίρους σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Πριν δώσω το λόγο λοιπόν στους προσκεκλημένους μα θα ήθελα να δώσω όμω την ευκαιρία στην κυρία Πασκάλη Κρουνή, την εισηγητριά μα, πολύ σύντομα να παρουσιάσει την, ε, το θέμα και στη συνέχεια κάθε ειδικό θα έχει περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή του. Κυρία Κρουνή, μπορώ να έχω 5 λεπτά πρόεδρε, 5 λεπτά μου δυνατά. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, τα δύο ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τι 7 Οκτωβρίου από την Ολομέλεια καταδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον των Ευρωβουλευτών για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το μέλλον τη πολιτική συνοχή Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένουν όμω ακριβή αρκετά ερωτηματικά και έτσι, διατυπώνω, έτσι τρέφω πολλέ ελπίδε από τι απαντήσει που ελπίζω ότι θα λάβουμε σήμερα από του εμπειρογνώμονε μα και τη συζήτηση που θα κάνουμε μαζί του, έτσι ώστε να μπορέσω κατά την προετοιμασία του εις προσεχούς εκθέσεως για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έχω αρκετά ο υλικό στη θέση μου ώστε να το λάβω υπόψη. Είναι καθήκον μας λοιπόν να προσδιορίσουμε αποτελεσματικά μέσα για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει ε, της ε, ε, πολιτικής 2020, 75% πλήρους απασχόληση από το 2020, που είναι πολύ φιλόδοξο στόχος και ασφαλώς θα πρέπει να δισκεδαστούν οι δυνάμεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι το πρώτο και το αρχαιότερο δημοσιονομικό μέσο για την ε, ενίσχυση της απασχόλησης στην Ευρώπη και έτσι θα πρέπει από νομοθετικής πλευράς να ενισχύσουμε την παρουσία μας ε, την ευρωπαϊκή αλλά και την ερατότητά του, γιατί όπως είπα δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε ένα εργαλείο στα χέρια μας, ένα μέσο στα χέρια μας το οποίο θα είναι αποτελεσματικό. Οργανώθηκε λοιπόν μια ομάδα εργασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με πρόεδρο την υποφαινομένη και έχουμε διαρκεί επαφέ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανταλλαγή απόψεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς το χρονοδιάγραμμα τώρα. Ποια είναι τα θέματα, τα γεγονότα, οι εξελίξεις στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Πριν από μερικού μήνες έδωσε μια, έκανε μια ακρόαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συμμετοχή τη Προέδρου και τη υποφαινομένη ε, για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είχαμε επίση το ψήφισμα για το ε, μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο Κοινοβούλιο με τους κατάλληλους, με τους κανόνες που προσδώσαμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που, είναι, που προσυδειάζουν στις ε, ιδιαιτερότητες του. Επίσης θα δημοσιευθεί η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, πολιτική συνοχή. Λυπούμε όμως γιατί δεν την έχουμε εγκαίρω στα χέρια μας, ώστε να μπορούσαμε να τη συζητήσουμε ήδη σήμερα. Και η θέση εφαρμογή βέβαια της συνθήκης Λισαβόνας ε, άλλαξε πολλά πράγματα και έτσι είναι συναρμόδια για λήψη αποφάσεων αρχή το Κοινοβούλιο, άρα απόσπαστο κομμάτι τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Επίση, η συζήτηση επί τη ουσία, όπω αντιλαμβάνεστε, πρέπει να αντέχει τη πλήρου ε, προσοχή μα. Έχουμε μια πρόταση νομοθετικών ε, κειμένων ε, που περιμένουμε περί τα μέσα του 2011 και μέχρι τότε πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, να παρακολουθούμε την κατάσταση και τι εξελίξει για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε αποτελεσματικά και ενεργά στι συζητήσει. Υπάρχουν και οι δημοσιονομικέ πτυχέ βεβαίω, η σημασία που θα αποδώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που του αρμόζει φυσικά, αλλά και η κατάλληλη πρικοδότηση που έχει τεράστια σημασία και άρα θα πρέπει ιδιαίτερη σημασία να αποδώσουμε στην προσοχή των ε, συναδέλφων της Επιτροπής ε, ΣΥΡ, έτσι ώστε να έχουμε αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ε, δύο επιτροπών. Όσον αφορά την επισκόπηση των δημοσιονομικών 19 Οκτωβρίου εφέτο, δεν μα επέτρεψε να προχωρήσουμε αρκετά γιατί δεν έχουμε στοιχεία οικονομικά στη θυσή μα, μόνο μία ένδειξη ενίσχυσης η οποία αναφέρεται στην κατάρτιση και την εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού. Ένα-δύο σημεία που είναι τα πιο σημαντικά θα ήθελα να φέρω κλείνοντας κυρίε και κύριοι. Πρώτα απ' όλα το ΕΚΤ είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Θα πρέπει να ενισχυθεί έτσι ώστε και να διαφυλάξει αυτές τις δραστηριότητες αλλά και να καταπολεμήσει τη φτώχεια και πάνω απ' όλα να φέρει τον πολίτη μέσα στην αγορά εργασίας, όχι άλλες λύσεις δηλαδή. Αυτή είναι, αυτό το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό αλλά και πιο απλό μέσω το ΕΚΤ. Δεν είναι, Δεν το δηλαδή μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσεως και με τόσο υψηλή οικονομία στην Ευρώπη, να μην αξιοποιούνται 100% τα οικονομικά μέσα του ΕΚΤ, άρα θα πρέπει και να εξορθολογήσουμε τις διαδικασίες που είναι αποθαρρυντικές μερικέ φορές για τους χρήστες και να ενισχύσουμε τα μέσα, ε, τα πρακτικά. Επίσης θα πρέπει το ΕΚΤ τρίτον να παραμείνει στην υπηρεσία κάθε περιφέρεια, στην ε, υπηρεσία της κοινωνική και οικονομικής συνοχής για κάθε περιφέρεια, που, εκ των οποίων ορισμένες έχουν φτώσει ανάγκε από κάποιε άλλες και γι' αυτό θα πρέπει να προσδοριστεί ένα πιο καλά προς προσαρμοσμένο ανάγκε των περιφερειών πλαίσιο και πάνω απ' όλα πλαίσιο προσαρμοσμένο στι ανάγκε των ανθρώπων. Και πέραν αυτού, οι θεσμικέ πτυχέ, η, αυτόμα... η αυτόνομη διαχείριση, η διαχείριση περιφέρεια θα πρέπει να διατηρηθούν έτσι ώστε πέραν του οικονομικού εντολέα να υπάρχει η δυνατότητα της απορρόφησης των κονδυλίων εκεί που είναι αναγκαία αυτά. Και τέταρτον, ε, θα πρέπει ο στόχος να είναι πάντοτε η καταπολέμηση του αποκλεισμού του κοινωνικού ή τη απόλυτη θέση εργασία. Τέταρτον, σε μια περίοδο οικονομική κρίσης. περιμένουμε πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί ένα, μια καλή οικονομική χρηματοδότηση, πρικοδότηση για το ΕΚΤ, αλλά μην λησμονούμε και τις ευθύνες των κρατών μελών, γιατί η Ευρώπη δεν έχει συσταθεί για να αναλαμβάνει κάθε είδους άχθος. Έτσι λοιπόν και όταν ε, αναφερόμαστε στις συνθήκες που το 1950 οδήγησαν τους ε, ε, προκατόχους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους προπάτορες να θεσπίσουν το Ευρωπαϊκό Κεντρικό Ταμείο, ε, πρέπει να διαρωτηθούμε αν οι ίδιες συνθήκες επικρατούν ακόμη και σε ποιο βαθμό χρειάζεται να το προσαρμόσουμε σε νέες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα παρακαλώ τους τρεις εμπειρογνώμονες μας να λάβουν το λόγο. Ο κύριος Κάρλος Τορτουέρο πρώτος, αρμόδιος στην Ισπανία για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Κύριε Τορτουέρο, έχετε δέκα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα καταρχά ε, να σας μεταφέρω τους θερμότερους χαιρετισμούς του κυρίου Φερνάντες, ο οποίος ε, η οποία, συγγνώμη, κυρία Φερνάντε, η οποία είναι υπεύθυνη ε, για όλα τα ζητήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ισπανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στη σημερινή ακρόαση για να συμβάλλω κι εγώ στην ε, συζήτηση αυτή για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να επενδύσει κανείς ε, στους ανθρώπους για να υπάρχει η Ευρώπη της ε, κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης. Είναι δύσκολες οι οικονομικές συνθήκες, βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης, αυτό σημαίνει ότι έχουν ακόμη μεγαλύτερες ανάγκες ε, ε, οι πολίτες μας, ώστε να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και να υπάρχει και ένα εργαλείο που μπορεί να τους διευκολύνει, ειδικά όσους θέλουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Εμείς έχουμε στην Ισπανία ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα ειδικότερα για τα ζητήματα κατάρτισης και απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική εμπειρία που μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε το μέλλον, λαμβάνοντα υπόψη ε, όλα όσα μα έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για την ισπανική εμπειρία και αυτή θα είναι και η συμβολή μου στη συζήτηση. Θα ήθελα να επιμείνω στη βελτίωση του ρόλου και της ορατότητας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, τη μείωση της φτώχειας, ανάπτυξη ε, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των υπηρεσιών απασχόλησης. Όλα αυτά πρέπει να είναι αντικείμενο μιας μόνιμης εξέλιξης και αναθεώρησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο ώστε να λάβουν χώρα οι απαραίτητες αλλαγές, λαμβάνοντας λαμβάνοντας υπόψη ε, την, ε, τις διαφορετικές ανάγκες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και σε άμεση ε, σχέση με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε να ενισχύσουμε κυρίως τα άτομα με τις περισσότερες ανάγκες, βελτιώνοντας την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές, ποιες είναι οι πλέον καινοτόμες πρακτικές που θα δώσουν τη δυνατότητα στις πολιτικές μας ε, να αποκτήσουν ε, νέα πνοή. Για παράδειγμα, η πολιτική ανθρωπίνων πόρων. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε περισσότερες ε, ε, καινοτομίε ε, στα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα και επίση να δούμε το θέμα τη διακυβέρνηση σε διάφορα επίπεδα. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η πολιτική διαχείρισης ε, ανθρώπινου δυναμικού είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και σε τοπικό επίπεδο. Είναι λοιπόν απαραίτητο να ε, συνεργαστούμε στην προσπάθειά μας αυτή με τους ε, τοπικούς μας εταίρους. Κάτι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ενθαρρύνουμε μία αίσθηση ε, πολιτικής πιο ενεργό, πιο απτή, βάσει των τοπικών συνθήκων και μάλιστα αξιοποιώντας τις εμπειρίες των ανθρώπων που δουλεύουν επί τόπου. Θέλουμε να συμπληρώσουμε τις προσπάθειες των εθνικών προγραμμάτων. Έχουμε Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και τις περιφερειακές αρχές οι οποίες εφαρμόζουν επιτόπου ε, τις ε, αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο με τη δέουσα ευελιξία και επίσης υπάρχει και το τοπικό επίπεδο που είναι το πιο κοντινό ε, στα, στους ενδιαφερομένους. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια προσέγγιση η οποία πηγαίνει και από κάτω προς τα πάνω αλλά και από πάνω προς τα κάτω να μην ε, ξεχνούμε ότι τα διάφορα προβλήματα είναι συνήθως πολύ περίπλοκα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να είναι σύνθετες και οι πολιτικές μας. Δεν είναι μόνο θέμα αναζήτησης εργασίας, είναι, υπάρχουν και ζητήματα στέγασης, εκπαίδευσης και υγείας. Πρέπει λοιπόν ε, να ε, δούμε τη συμπληρωματικότητα με ένα ακόμη διαρθρωτικό ταμείο για την ανάπτυξη των περιφερειών που είναι το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δεν πρόκειται βέβαια να... Ε, συγχωνευτούν τα δύο ταμεία, έχουν δύο διαφορετικούς ρόλους, όμως μπορούν να δρουν συμπληρωματικά. Με αυτονομία το καθένα, αναπτύσσοντας κοινά προγράμματα όποτε χρειάζεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Προσαρμογής ε, στην Παγκοσμιοποίηση και με τα άλλα ε, εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι, υπάρχει συμπληρωματικότητα ε, στη θεωρία, αλλά πρέπει και οι διάφορες δράσεις να είναι συμπληρωματικές. Επίσης πρέπει να βελτιώσουμε την ορατότητά μας. Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι ένα ταμείο που βοήθησε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο λίγο γνωστό στους Ευρωπαίους πολίτες. Εμείς έχουμε, μια προσπάθεια, έχουμε κάνει μια προσπάθεια ενημέρωση στην Ισπανία και σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο είμαστε η τρίτη χώρα για την οποία η ορατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι ε, υψηλότεροι. Οι Ισπανοί πολίτες γνωρίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τους στόχους του και αυτό βέβαια δεν μας εμποδίζει από το να προσπαθούμε να ε, ε, ενισχύουμε όλο και περισσότερο τις προσπάθειές μας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να συμπληρώσουμε και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ισπανία αυτό σημαίνει αξιολόγηση των υπηρεσιών ε, του Ταμείου στις κοινωνίες μας και ειδικότερα για τα άτομα που βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση. Επίσης θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα ελέγχου που θα βασίζεται στα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή η διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία, από ε, διοξοδικούς ελέγχους που εξασφαλίζουν ότι τα ε, διαθέσιμα ποσά ε, αξιοποιούνται με πλήρη διαφάνεια. Όμως δεν πρέπει να παραλύουν και όλα στα επιχειρησιακά προγράμματα που είναι επωφελή για χιλιάδες άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου, αλλά διαδικασίες ελέγχου που δεν ε, καταπνίγουν τελικά το σύστημα. Θέλουμε λοιπόν κανόνες παιχνιδιού σαφείς, απλούς, ε, χωρίς να υπάρχει αντίφαση με μία ενιαία πηγή πληροφοριών που διευκολύνει και τη διαχείριση και τον έλεγχο. Είναι λοιπόν ε, αδιαμφισβήτητο ότι σε αντίθεση με άλλα ταμεία, ο αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι δυσκολότερο να προσμετρηθεί και είναι δύσκολο να τον, να τον γνωστοποιήσουμε ε, στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Γι' αυτό ακριβώ χρειαζόμαστε και εργαλεία αξιολόγηση του αντικτύπου αυτού πρέπει να είναι ε, καλύτερη η παρακολούθηση των ε, δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ώστε να είναι σαφέστερες οι ευθύνες. Όταν οι στόχοι ε, επιτυγχάνονται, πρέπει αυτό να είναι μετρήσιμο και να το γνωρίζουν όλοι και όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο. Είναι σημαντικό οι επιδοτήσεις να φτάνουν όσο το, το, το δυνατόν συντομότερο σε όσους τις χρειάζονται. Πρέπει δηλαδή να ε, ε, έχουμε μέτρα βελιξίας ε, και απλοποίησης, όπως επίσης και μικρότερη διάρκεια προθεσμιών πληρωμών. Πώς είναι δυνατόν τώρα να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, πώς γίνεται η συντονισμός με τους κοινωνικούς εταίρους. Σε εθνικό περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται μέσω δικτύωσης η προσπάθεια αυτή, δηλαδή συνδέουμε την απασχόληση με την ε, ενσωμάτωση. Στην Ισπανία πάντοτε δίναμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτού του είδους τη συνεργασία και στην αύξηση της συμμετοχής των κοινωνικών ε, παραγόντων, των ε, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και των οργανισμών κοινωνίας των πολιτών για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ε, χάρη στην ε, ε, διακρατική συνεργασία, μπορούμε από κοινού να αναζητήσουμε, προβλήματα, να αναζητήσουμε λύσεις στα προβλήματα που είναι κοινά για όλα τα κράτη-μέλη. Ένα πολύ απλό παράδειγμα το δίκτυο που δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του πληθυσμού των Ρωμά στην Ευρώπη εμείς θεωρούμε ότι η ισπανική εμπειρία ε, στέφθηκε με επιτυχία και ότι μπορούμε να ε, αποτελέσουμε παράδειγμα ε, για αντίστοιχες προσπάθειες σε άλλα κράτη-μέλη. Είδου λοιπόν κάποιες ιδέες για το μέλλον. Έχουμε πολύ σημαντική εμπειρία και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού διαφόρων ομάδων Έχουμε εμπειρογνώμονε επιτόπου που γνωρίζουν πολύ καλά τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι ομάδε αυτέ. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ειδικότερα τα άτομα με μεγαλύτερες δυσκολίες και προσπαθούμε επίσης να ενσωματώσουμε τη διάσταση της ισότητας των φύλων που πάντοτε γινόταν σεβαστή στην Ισπανία και εξακολουθούμε να την προωθούμε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτούς τους μηχανισμούς mainstreaming να ε, συνεχίσουμε να τους ε, προωθούμε σε, ευρωπαϊκό, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε επίπεδο Εθνικών ε, Κοινοβουλίων, τοπικών αρχών. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ φιλόδοξα πολύ φιλόδοξους στόχους, περισσότερη συνεργασία για να μπορέσουμε να κάνουμε συγκριτική αξιολόγηση ε, με τους διάφορους βέβαια ε, προσανατολισμούς ε, επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχει θέσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κρίση και η ανεργία Ε, δείχνουν ακόμη περισσότερο την ε, σημασία της, ε, του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Ταμείου. Η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 ε, έχει θέσει κάποιους στόχους ε, και επομένως θα είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Θα πρέπει να δούμε που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να τους βοηθήσει και αυτό για να γίνει χρειάζεται μεγαλύτερη ορατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων και καλύτερο συντονισμό με παράλληλη απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια με σεβασμό των ε, οικονομικών περιορισμών. Χρειαζόμαστε ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως σας είπα και προηγουμένως, με ε, διενέργεια ελέγχων, αλλά δεν είναι ο οικονομικό έλεγχο ο αποφασιστικό. Ο αποφασιστικό είναι ο τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βοηθά του πολίτε. Είναι πραγματικά κατάλληλο το είδο τη βοήθεια. Μπορούμε πάντοτε να τη βελτιώσουμε. Γιατί όσο καλύτερα, ε, όσο βελτιώνουμε τι προσπάθειέ μα, ε, τόσο πιο ορατό γίνεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σα να σα ενισχύσω σε οποιαδήποτε προσπάθειά σα. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον κύριο Μάρκ Γκαρσέ, ο οποίος είναι και γενικός γραμματέας των διαφόρων ενώσεων, στις οποίες συμμετείχατε και Γκαρσέ, για την επαγγελματική αποκατάσταση και καθοδήγηση και είστε και συγγραφέας πολλών έργων, συγγραμμάτων και άρθρων που μπορούν να μα διαφωτίσουν για τη λειτουργία και το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτήν την παρουσίασή σας. Ταπεινοφρόνος θα ήθελα να σα κάνω κάποιε προτάσει και με κάθε επίση ταπεινότητα να τι υποβάλω στα μέλη του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να αναπτύξω πέντε σημεία στην παρουσίασή μου. Καταρχάς, ξεκινώντας από το τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προχωρώντας μετά στο πώς θα, αλλάξουν, ε, πώς θα αλλάξει το τοπίο το 2020, βλέποντας το σταυροδρόμιο το 2008-2009 με την κρίση με, που πλήττει την απασχόληση, αυξάνει την ανηλικία, αλλάζει την εθνική και την κουλτούρα και το ρόλο των τραπεζών ως κινητηρίου δυνάμεις της οικονομίας. Μια νέα λοιπόν κουλτούρα, μια νέα νοοτροπία με έλλειψη εμπιστοσύνη, έλλειψη ιδεολογιών ε, σε σχέση με αυτή την μεγάλη πρόκληση της Ευρώπης, το μεγάλο ευρωπαϊκό ιδεώδες. Πρέπει λοιπόν η λειτουργική προβολή του ΕΚΤ να προαχθεί και αυτό είναι μια σοβαρή πολιτική προτεραιότητα. Υπάρχει ανάγκη για ισχυρές δηλώσεις, ισχυρές τοποθετήσεις, όπως η δήλωση της Λισαβόνας ε, τον καιρό που έγινε. Ή θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να συσχετιστεί με ένα κατάλογο προτεραιοτήτων για την οικοδόμηση της κοινωνικής Ευρώπης με κάποιο υπόβαθρο ευρωπαϊκών κοινωνικών δικαιωμάτων που να είναι αρκετά λογικά Ίσως η δήλωσή μου αυτή να είναι προκλητική, όμως κάτι τέτοιο θα ήταν ένα βήμα προόδου, ένα βήμα μπροστά. Πρέπει λοιπόν να διευρυνθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και το πεδίο δράσης του. Έχουμε το ΕΚΤ, το οποίο μπορεί μέσω των καταρτήσεων που προσφέρει, των σχηματισμών του μάλλον, συγγνώμη, να επιτρέψει ανάληψη πρωτοβουλίας και προσωπική ανάληψη ευθύνης. Η νοοτροπία του επιχειρήν, τα αποτελέσματα των εγχειρημάτων, η προσωπική δράση. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη μια νέα εκπαίδευση. Πρέπει το άτομο να γίνει υπεύθυνο και να παίρνει στα χέρια την ίδια του τη μοίρα. Μια άλλη διάσταση που πρέπει να προσφέρουμε στην κατάρτιση είναι η έρευνα και η καλλιέργεια των νέων μοντέλων για τι επιχειρήσει όπω το coaching, η εναλλαγή μεταξύ πρακτικής και του ε, e-learning, ε, η κοινωνική διάσταση και η οικονομική, προκειμένου να διασφαλιστεί ταυτόχρονα και η νοητική υγεία, μια τρίτη πρόταση, θα μπορούσε να είναι να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση εντός επιχείρησης, με ε, μια θέση εργασίας στο τέλος, στο χέρι. Επιτά πρέπει να δώσουμε αξία και στα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά και στα υψηλότερα, εκεί που έχουμε νέες τεχνολογίες. Επίσης, μια πρόταση εισαγωγής της επαναπροσαρμογής ε, στο ψυχοκοινωνικό επίπεδο προς την απασχόληση και για πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Γιατί, γιατί διαπιστώνουμε ότι το κοινό έχει καταληφθεί από ένα σύνδρομο πρόορη συνταξιοδότηση ε, από μια ηλικία και μετά. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ε, θα μας ε, πούν ότι είναι καλύτερο να βγαίνει κανείς νωρίτερα στη σύνταξη, τέτοια δικαιώματα θα επιδιώξουν. Εκεί λοιπόν βλέπουμε πολλούς ανθρώπους αυτή την ε, νεαρή ηλικία να παθαίνουν κάποιο είδους κατάθλιψη γιατί η δυνατότητα για να εργαστούν υπάρχει ακόμη. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να εξεύρουμε μια νέα μορφή επαναπροσαρμογής επαγγελματικής ώστε να αλλάξει επαγγελματική μοίρα, πορεία των ανθρώπων αυτών και κοινωνική τους ένταξη. Εδώ υπάρχει ένας νέος τομέας που πρέπει να διερευνήσουμε. Επίσης, η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να επιτρέπει και την δημιουργία απασχόλησης μερικές προτάσεις. Κατά πρώτον, η δημιουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να προσφέρει και οικιακές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες εγκύτητας στην κοινότητα. Εδώ μιλάμε για μία πασαρέλα, ένα πέρασμα που πρέπει την αξιοποίηση του κοινού, ιδίως για πολίτες που έχουν περάσει από περιόδους τελμάτωσης, αδράνειας. Δεύτερη πρόταση, η δημιουργία συστημάτων διαρκούς παροχής υπηρεσιών, ε, συνδυασμένα με μια πολιτική κοινωνική συνοχής. Εδώ προσπαθώ να κάνω παραλληλισμό μεταξύ ΕΚΤ και κοινωνικής συνοχής, τοπικής συνοχής. Τρίτη πρόταση, ε, κάπως πιο προκλητική ακόμη, να, ε, να επινοήσουμε ή να προτείνουμε την κοινωνική επιχείρηση γενικού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερο νομικό καθεστώς κάπως με το πρότυπο των ε, ήδη υπαρχόντων εταιριών. Γιατί, γιατί η στόχευση της ενεργείας, ένα συγκεκριμένο κοινό, είναι παρόμοιο σε όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη. Εγώ ταξίδεψα παντού με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και το αντιληφθήκαμε ξεκάθαρα αυτό. Τα προβλήματα που έχουμε στη δική μας χώρα είναι παρόμοια με αυτά που έχουμε στις άλλες στην Πολωνία, τη Βουλγαρία και το καθεξής. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε μια νέα μορφή κοινωνικής επιχείρησης. Το ΕΚΤ και το ΦΕΝΤΕΡ θα μπορούσαν να συνδυάσουν ε, τις, ε, τα κονδύλια για αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Επίση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να ασχοληθεί με τι τοπικέ κοινότητε και τι περιφερειακέ με κυβερνητικέ οργανώσει, διότι είναι κατεξοχήν ε, συνεργάτε για να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση σε κοινωνικέ εταιρείε ε, δημοσίου ενδιαφέροντο. Η κοινωνική λοιπόν εταιρεία με συγκεκριμένο νομικό καθεστώ θα έχει και περιφερειακή διάσταση. Τέταρτη ιδέα, να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ. Αυτό προφανώς είναι περισσότερο μια διατομιακή προτεραιότητα. Στην επιχείρηση όπου εργάζομαι εγώ έχουμε επινοήσει και δημιουργήσει την έννοια της κοινωνικής αποδοτικότητας εντός ε, εισαγωγικών, ε, κοινωνικής κερδοφορίας. Αυτή η έννοια θα μπορούσε να διακριθεί από την ε, κοινωνική διάσταση την απλή. Εδώ η κοινωνική κερδοφορία μιλάμε έχουμε μια ανάλυση, μια μελέτη ετήσια με λεπτομέρειες και συγκεκριμένε κατηγορίε και καταλόγου για τι υπηρεσίε που προσφέρονται στην κοινωνία και στι κοινότητε τι τοπικέ. Όπω είπε και προλαλή σα, δεν χρειάζεται να κοιτάμε μόνο του οικονομικού δείκτε, δεν αρκεί μάλλον αυτό. Αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και του δείκτε για τι κοινωνικέ διαστάσει, όπω η κοινωνική χρησιμότητα, η ευστοχία και το τι προσφέρεται, η αξία, η αλληλεγγύη, η αξιοποίηση του τελικού αποτελέσματος σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά θα φροντίσουν να συμπυκνωθούν σε ένα σύγγραμμα που ονομάζεται η οικονομία δεν μπορεί να είναι μόνο κοινωνική, θαυμαστικό. Εδώ λοιπόν χρειάζονται διαδικασίες που να στηρίζονται οικονομικώς από τα κράτη μέσω του ΕΚΤ. Η καλή διακυβέρνηση του το τομέα της οικονομίας των υπηρεσιών, των συλλογικών υπηρεσιών, πρέπει να διέπεται από κανόνες που το έκτο μπορεί να προάγει. Η καλή διακυβέρνηση στο κοινωνικό επίπεδο μπορεί να δώσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο κοινό, να αποδείξει ότι έχει καλές επιδόσεις η Ευρώπη, δίνει αποτελέσματα και στους ίδιους τους πολίτες, απευθείας στους πολίτες. Πέμπτη παρατήρηση. Λίγα λόγια για το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Η κοινωνική εταίροι είναι οι συνεργάτε μα από την πλευρά των πολιτών. Το Κοινοβούλιο είναι μια μορφή έκφραση ακριβώ τη βούληση των πολιτών. Υπάρχουν και μη κυβερνητικέ οργανώσει και ενώσει πολιτών που όμω δεν εκπροσωπούνται με ίσο τρόπο, ισότιμα. Υπάρχει μια διάσταση όμω εδώ ενωσιακή συλλόγου που ε, προάγει τα κοινωνικο-οικονομικά συμφέροντα. Το Ταμείο λοιπόν θα μπορούσε να έχει διευρυμένο ρόλο. Θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτεροι και πιο στενοί συσχετισμοί μεταξύ των ε, κοινωνικών ενώσεων και του ΕΚΤ. Προτείνουμε επίσης η κοινωνία των πολιτών, η οποία εκπροσωπείται από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και η οποία συχνά καλύτερα να λάβει δράση στο τοπικό επίπεδο, να εκπροσωπείται και στο ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω φόρουμ, συγκεκριμένων φόρουμ, γενικών για τι ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει που ασχολούνται με τη λειτουργία του ΕΚΤ. Αυτή η πρόταση πιστεύουμε ότι είναι ενδιαφέρουσα στο βαθμό όπου έχουμε μια σταδιακή επαναδίπλωση των κρατών ε, στον εαυτό τους. Ε, θα μπορούσε λοιπόν ένα φόρουμ να συμπληρώνει τις δράσεις του ΕΚΤ ή να απευθύνεται απευθείας στο ΕΚΤ. Τι θα έδινε ως σε ένα τέτοιο φόρουμ των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα έδειχνε τις διακυμάνσεις, τις τάσεις και τη γενικά φαινόμενα της κοινωνικής διάστασης. Θα ήταν ένα εργαστήριο που θα αναλύονται κοινωνικές γνώσεις και τα κοινωνικά διδάγματα όπως τα βλέπουν όσοι δρούν στην πράξη. Και θα μπορούσε να εξεύρει τα συστατικά μιας κοινωνικής νοοτροπίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Τα συστατικά αυτά, το έχουμε υπογραμμίσει επανειλημμένως, έχουν την εξή έννοια. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν είναι διακρατικό. Θα πρέπει το διακρατικό χαρακτήρα να το αναζητήσουμε σε άλλα εγχειρήματα. Δεν θα ήταν άστοχο να προσθέσουμε εδώ στοιχεία όμως διατομιακά και διακρατικά ακριβώς στα εθνικά ταμεία ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά. Ξέρουμε ότι η γεωγραφική φραγμή είναι στο μέσο που πειραματιζόμαστε για τις ανταλλαγές μας μέσα από τον φόρουμ. Είναι προφανές ότι η κρίση μας οδηγεί σε ριζοσπαστικοποίηση των θεσεών μας. Περισσότερος φιλελευθερισμός, περισσότερη συνδικαλιστική δράση. Πρέπει να αναζητήσουμε μια μέση οδό. Μια κοινωνική χάρτα η οποία να συμφιλιώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα εργασιακά των πολιτών και τις ευθύνες που υπάρχουν γύρω από αυτά τα δικαιώματα. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να παρέμεινα στα όρια του χρόνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτές τις ιδέες που μας δώσατε και για τις πρόπτικες για το μέλλον, δεδομένες της πείρας σας σε αυτόν τον τομέα, που είναι σημαντική. Δίνουμε το λόγο στον τρίτο μας ομιλητή, είναι Ούγγρος, ο κύριος Ιστφανταντέ. Είστε σύμβουλος του δικτύου της Ουγγαρίας για την καταπολέμηση της ένδυας, ιδίως ό,τι σχετίζεται με τα διευθυντικά ταμεία. Έχετε το λόγο και εσείς για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που παίρνω το λόγο. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Είναι βέβαια αδύνατο να συνοψίσει κανείς ε, σε 10 λεπτά ένα τόσο μεγάλο θέμα. Και όταν έπρεπε να προετοιμαστώ για την παρουσίαση αυτή, πραγματικά προβληματίστηκα γιατί σκεφτόμουν πολλή ώρα σε ποιο θέμα θα έπρεπε να δώσω προτεραιότητα, ποιος είναι ο κοινό παρονομαστής που θα μπορούσαμε να έχουμε σε μια τέτοιου είδου συζήτηση. Και θα έλεγα ότι είναι ο ρόλος της αγοράς εργασίας. Αυτός είναι ο σημαντικότερος ρόλος. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τα καλύτερα μέσα εδώ στην Ευρώπη να βρει ο καθένα θέση του στην αγορά εργασία. Και τότε πρέπει να διαρωτηθούμε και τι είδου Ευρώπη θέλουμε. Τι ζητούμε από την Ευρώπη. Ή σε τι θα πρέπει να ε, επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας για να υπογραμμίσουμε τα σημεία που αποτελούν πλεονέκτημα, που είναι τα ε, σημεία στα οποία έχουμε περισσότερες ικανότητες και που θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη υποστήριξη. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε πάντα για πρόσωπα, για ανθρώπους και αυτούς πρέπει να βλέπουμε πάντα στη θέση τους, σε μια θέση εργασίας και όχι όργανα ή φορείς απρόσωπους. Πού λοιπόν θα αναστήσουμε τους δείκτες, πού θα επιδείξουμε αποτελεσματικότητα, πόσο θα προσμετρήσουμε τις δεξιότητες και τον αριθμό των κατερτισμένων και εξειδικευμένων εργαζομένων. Και πόσο μπορεί να υπολογιστεί η απασχολησιμότητα των ανθρώπων αυτών. Επίσης, σε ποιο σημείο θα πρέπει να υπολογιστεί αυτή η απασχολησιμότητα. Δεν είναι νομίζω τώρα η στιγμή να την συζητήσουμε σε εποχή οικονομικής κρίσης. Θα έπρεπε αυτό το θέμα να μας έχει απασχολήσει πολύ καιρό πριν. Και εν τέλει υπάρχει κάποιο είδους συνάντηση συνύπαρξη της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, των ανθρώπινων δυνατοτήτων και υπάρχει και ένα σημείο ε, που μπορεί να εξηγήσει, μια άποψη μπορεί να εξηγήσει σε ποιο σημείο της ζωής του ανθρώπου, σε ποιο χρονικό σημείο, σε ποια ηλικία θα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερα κονδύλια. Ε, λέμε παραδείγματι ε, ότι τα πρώτα πέντε χρόνια του παιδιού είναι κρίσιμα για να ε, μπουν τα θεμέλια της αγοράς εργασίας. Όσο πιο πολλές ε, υπηρεσίες μπορέσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά αυτά, στις οικογένειες αυτές που έχουν ανήλικα παιδιά, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η αναζήτηση από τα παιδιά αυτά μιας ε, θέσης στην αγορά Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, κάνουμε διαχωρισμούς και να επιλέγουμε ορισμένους μόνο ή επιφερειπίν μόνο τους φτωχές οικογένειες. Όλοι θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες. και εκείνοι οι οποίοι έχουν ε, ε, κάποια μόνιμη ασθένεια και οι πληθυσμοί των ε, Ρωμά και θα πρέπει όλες οι υπηρεσίες και το ΕΚΤ βέβαια να συνεργαστούν στενά. Τι απαιτείται λοιπόν. Ξέρετε ότι υπάρχει το σύστημα Atkinson που είναι γνωστό. Και ως προς την ε, διακυβέρνηση σε κάθε επίπεδο, οπουδήποτε έχουμε να κάνουμε με τον πολίτη, πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να πεμπολούμε ευθύνες λέγοντας ότι κάποιος άλλος έχει την αρμοδιότητα να ασχοληθεί με τους ε, πολίτες ή με τις ανάγκες των πολιτών. Και φυσικά δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι πάντοτε τα θεσμικά όργανα θα είναι εκείνα τα οποία θα ασχολούνται με το θέμα αυτό. Διότι αν περιοριστούμε στα θεσμικά όργανα και εξαντληθούν εκεί οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις, σε επίπεδο πολίτη δεν θα φτάνει πια τίποτα. Σας δίνω σαν παράδειγμα έναν κύβο δυσδιάστατο που μας δείχνει ότι αν θελήσουμε να ασχοληθούμε τους πιο ευάλωτους, με τις πιο ευάλωτες ε, ομάδες, θα πρέπει να κοιτάξουμε και τους δείκτες, αλλά και τις πολιτικές. Ιδάλλως θα μένουν πολλά κενά μέσα στους ε, κύβους. Όσον αφορά τις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα πρέπει να γνωρίσουμε ποιος είναι ο πάροχος, ποιος αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά. Στις μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν λέμε να προσφέρονται προς τρακονδύλια γιατί έχουν προσθέσεις ανάγκες, αλλά γιατί ξέρουμε ότι ο προϋπολογισμός ενός κράτους δεν μπορεί παρά να συμπληρώσει τους πόρου των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δεν αρκούν ώστε να εξασφαλιστεί η θέση εργασία για τους πολίτες, έτσι ώστε να υπάρξουν να υπάρξει υπαρκή υποστήριξη για συστήματα τη μια τέσσερα εργασία. Οι κυβερνητικέ οργανώσει, δηλαδή εκείνε οι οποίε ανεπίσημα αναπτύσσουν τη δραστηριότητά του και έχουν διαρκή επαφή με τον πολίτη σε καθημερινή βάση, σε βάση βοήθεια καθημερινή που του προσφέρουν, θα πρέπει να έχουν εν τέλει αρκετό δυναμικό και υποστήριξη θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική γιατί ακριβώς αυτή η ενίσχυση, αυτή η αρρωγή έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Και αν κοιτάξουμε τον αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε βεβαίως να προβούμε σε μία ε, αξιολόγηση, αλλά αυτό αν κοιτάξουμε τι είδους συστήματα υπάρχουν στα κράτη-μέλη και δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στην ε, φορολογική πολιτική και να αποκόψουμε την ε, ενίσχυση από το Ταμείο. Γιατί αν το πράξουμε αυτό, τα αποτελέσματα δεν θα είναι ποτέ ικανοποιητικά. Το μήνυμα νομίζω που αποστέλουμε είναι απλό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κονδυλίων με συμμετοχή στο μέγιστο των ε, φορέων, των ε, ε, οργάνων, των θεσμικών οργάνων μέχρι το τελικό στάδιο της ε, υλοποίησης και πάνω απ' όλα να γνωρίσουμε τι θέλουμε και όχι μόνο τι έχουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευχαριστώ για άλλη μια φορά το δίκτυο για την ε, καταπολέμηση της ένδυας, κυρίως των παιδιών, που μου επέτρεψε να εργαστώ στην υπηρεσία τους επί πέντε χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν και μετά θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε. Κύριο Στάρτον και μετά ε, κυρία Σρέτερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες ε, που μας μετέφεραν τις εμπειρίες τους ε, επιτόπου και για τον ε, ενθουσιασμό τους, για την πίστη τους στο Ευρωπαϊκό Κεντρικό, ε, Κοινωνικό Ταμείο όπως επίσης και στην, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Κάτι το οποίο εντάξει μου φαίνεται ένας ε, προφανής στόχος, αλλά μας βρίσκει και απολύτω σύμφωνος. Δύο σημεία θα ήθελα να θέσω, που αφορούν κυρίως τον προϋπολογισμό μας. Καταρχάς, το θέμα του μέλλοντος του πολιετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού και μέσω της, και μάλιστα, ε, μέσω της ειδική επιτροπής που συστάθηκε για αυτό το λόγο, όπως επίσης και για όλο το θέμα του προϋπολογισμού για το 2011, η οποία αφορά ένα πιο μακροχρόνιο προγραμματισμό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, αυτού του προγραμματισμού του πολιετού. Τι χρειαζόμαστε, πέντε χρόνια, επτά χρόνια, δύο φορές επί πέντε χρόνια. Τι ακριβώς ε, όλο αυτό το ζήτημα της, του πολιετούς προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων είναι ένα ζήτημα που τίθεται και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη από αυτού. Επίσης ήθελα να σας ρωτήσω και ποια είναι και η αίσθησή σας ε, επιτόπου αυτού του πολυετούς προγραμματισμού. Πώς το ζείτε εσείς καθημερινά. Ποια είναι η άποψή σας ε, και το λέω αυτό σε σχέση με αυτά που είπαν οι εμπειρογνώμονες σε σχέση με το πόσο βαριά είναι η διαδικασία ε, ελέγχου. Ένα ακόμη ζήτημα είναι αυτό της ε, συμπληρωματικότητας ε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου, του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Αν Αν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ε, κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να λέμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ήταν λιγότερο επιτυχές στο στόχο του. Ποια ακριβώς λοιπόν είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο ταμείων. Είναι διαφορετική η χρήση, η αξιοποίηση των κάθε, του κάθε ταμείου, το ένα εκ των υστέρων, το άλλο εκ των προτέρων. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε και εσείς τη δική σας άποψη για το θέμα αυτή της συμπληρωματικότητας μεταξύ αυτών των δύο ταμείων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σρέτερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περίπλοκο το θέμα. Και θα ήθελα μόνο να θέσω κάποια ζητήματα μετά όσα ακούσαμε. Φαντάζομαι ότι και στην πορεία της ομάδας εργασίας και στην Επιτροπή μας θα κληθούμε να εξετάσουμε εις βάθος τους μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ως προς τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και το δεδομένο ότι το ΕΚΤ δεν επιδρά πάνω σε μια περιφέρεια αλλά σε πρόσωπα, σε άτομα και αυτή είναι η στρατηγική του επιλογή. Τι λοιπόν ένα ερώτημα αναγκαστικά ως προς το μέλος των Ισοτικών Ταμείων μάλλον δύο ερωτήματα, αφενός με το ότι μέχρι τώρα δεν δόθηκε επαρκής προσοχή στο ότι υποχωρεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα κράτη-μέλη. Ε, έναντι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Πράγμα όμως το οποίο σημαίνει τελικά δεν εξυπηρετούν οι στόχοι που, είχε αρχικά, που είχαν αρχικά οριστεί για το έκτο. Και η δεύτερη ερώτηση, σε σχέση και σε συνδυασμό και με άλλα ε, ταμεία, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης περισσότερο, θα έλεγα, θα σήμερα ενδεχομένως ε, συνεργασ... συνδυασμένη χρήση των ταμείων έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η ε, λειτουργία τους. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων. Καλύτερα είναι κατακαιρματισμένο το έργο των Υπουργείων και έτσι δεν υπάρχει αυτή η συνεργατική δράση. Τι θα μπορούσε να γίνει λοιπόν κατά την άποψή σας έτσι ώστε να μην χρειάζεται να υποβάλλετε διπλή αίτηση σε δύο υπουργεία κτλ. όταν ε, ζητά κανείς υποστήριξη. Επίσης ένα ζήτημα το οποίο δεν ε, φύγει ικανοποιητικά είναι αυτό του gender budgeting, δηλαδή του προπολογισμού του στηριζόμενου στην υποστήριξη των φίλων. Αυτό προβλέπεται στον κανονισμό του ΕΚΤ. Δεν είπατε όμως αν πράγματι εφαρμόζεται. Επίσης, η κοινοτική πρωτοβουλία Equal. Αν δείτε στην αιτιολογική μας σκέψη υπαριθμών 6, υπάρχει αυτή η απέτηση από πλευρά του Κοινοβουλίου, την οποία μας δεν αξιοποιούν τα κράτη-μέλη. Σφάλμα μοιραίο για μένα. γιατί βλέπουμε ότι και στα μέτρα και στις ομάδες στόχου, αλλά και στο, στην περιγραφή των σχεδίων, υπάρχει η ανάγκη για το equal. Είναι ένας αγώνας στον οποίο έχουμε αποδεθεί εμεί από πλευρά του Κοινοβουλίου εδώ και πολύ καιρό και τα καταφέραμε, αλλά δυστυχώ δεν εφαρμόζεται. Και ευχαριστώ προκειμένου και τους τρεις ομιλητέ για τις παρατηρήσεις τους. Για δε το άρθρο 5, την περίφημη ρήτρα για τις μη κυβερνητικές οργανώσει. Έχουμε αγωνιστεί και για αυτό το θέμα, όχι με τόση επιτυχία όσο θα θέλαμε. Πάντως, καταλήγουμε τελικά ότι η, στο ότι η δομή των μη κυβερνητικών οργανώσεων έχει γίνει πιο επαγγελματική, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι καλά κάναμε και στήσαμε τη ρήτρα αυτή, καλά κάνει και υπάρχει η ρήτρα αυτή, διότι χάρη σε αυτήν πιστεύω συμβάλλουμε στην βελτίωση της ε, αποτελεσματικότητας τους και αυτό ακούω και από τα όσα είπε ο εκπρόσωπος του δικτύου ε, για την καταπολέμηση της φτώχειας που μας μίλησε για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και το σημαντικό τους ρόλο. Όμως από τους τρεις ομιλητές δεν άκουσα σχόλια για το πόσο αποτελεσματική η καινοτόμα είναι η προσέγγιση της διοίκησης, της δημόσιας διοίκησης στην υπόθεση αυτή. Γιατί στο παρελθόν είχαμε ταμεία τα οποία προωθούσαν την καινοτομία. Εν τω μεταξύ όμως φάνηκε ότι ήταν πολύ γραφειοκρατικές οι δομές τους, καταργήθηκαν. Δεν έχουμε όμως αντίστοιχες, ε, αντίστοιχες δομές που να τα αντικαθιστούν. Πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα έτσι, αρκούν ή όχι. Ε, για δε το Ταμείο για την Προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, στην θα ήθελα να σημειώσω ότι διαφωνώ πλήρως με τον προλαλήσαντα. Είναι για μένα πολύ καλύτερη η ε, δράση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που προσπαθεί να προλάβει τις εξελίξεις ε, και γι' αυτό το προτιμώ στο Ταμείο για την προσαρμογή στην πίση. Κύριε Πρόεδρος, ευχαριστώ και παρακαλώ τους συναδέλφους να συντομεύουν, διαφορετικά θα προλάβουμε να δώσουμε το λόγο στους ειδικούς μας. Και αν είναι έτσι, δεν υπάρχει λόγος να τους θέτουμε ερωτήσει. Ο κύριος Σωρή και μετά ο κύριος Κομφεράτη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω κι εγώ ότι χάρηκα πολύ που άκουσα αυτήν την προσέγγιση από πλευράς εμπειρογνωμόνων, δηλαδή ότι η συμμετοχή στην αγορά εργασίας ε, αποτελεί το επίκεντρο των προγραμμάτων και ε, το επίκεντρο του νέου προγράμματος ε, εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Και θα ήθελα μάλιστα να πω ότι είμαστε τυχεροί γιατί οι οι ιδέες ε, για τη στρατηγική, τα θέματα της διακυβέρνησης, ε, οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν την διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέτουν τα ίδια ερωτήματα. Μετά από πολλά χρόνια απογοήτευσης και έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης, βλέπουμε επιτέλους ότι η οικονομική πολιτική και η κοινωνική πολιτική σιγά σιγά αρχίζουν να συγκλίνουν. Και επίσης θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε καλύτερα την ευκαιρία αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πει πολλάκις ότι θα έπρεπε να βοηθήσουμε όσους ζουν σε συνθήκες φτώχειας, να ε, βελτιώσουν την κατάστασή τους. Τα παιδιά των ανθρώπων αυτών, αν ε, βελτιώσουμε την κατάστασή τους τώρα, θα έχουν καλύτερες ε, προοπτικές για το μέλλον. Όσον αφορά τώρα τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, έχουμε ακόμη πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Καταρχάς πρέπει να βελτιώσουμε τους δείκτες νομίζω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε τους τομείς στους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και επίσης πρέπει να αναλύσουμε κατά πόσο η αξιοποίηση των πόρων αυτών ε, έχει αποτέλεσμα ή όχι. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε δείκτες, επαναλαμβάνω. Ακούσαμε ότι κάποια προγράμματα στέφθηκαν με επιτυχία. Πώς το γνωρίζουμε αυτό, εγώ θα ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση. Ε, πώς το μετράμε αυτό, έχουν δημιουργηθεί θέσεις απασχόλησης, ε, υπήρξαν περισσότεροι φοιτητές ε, στο πανεπιστήμιο ή μαθητές στο σχολείο, περισσότεροι άνθρωποι είχαν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ήταν λιγότερο επισφαλής οι θέσεις απασχόλησης. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένους στόχους καταρχάς και μετά να έχουμε και τους απαραίτητους δείκτες για να καταλάβουμε εάν καταφέραμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς ή όχι. Όλα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορούμε να... Ε, να μπορεί να λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σωστά. Επίσης, συνδυασμός των θεμάτων εκπαίδευσης Τη απασχόλησης και πολλών άλλων πτυχών. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν δεν υπάρχει συντονισμός με τα διάφορα εθνικά προγράμματα ή και διεθνή προγράμματα που σκοπό έχουν να επιτύχουν τους ίδιους στόχους. Θα ήθελα μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες για την παρουσία τους και για την παρουσίαση των ιδεών τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κομφεράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου φαίνεται ότι είναι διαδεδομένη άποψη ότι η υλοποίηση των στόχων είτε οικονομικού χαρακτήρα είτε κοινωνικού χαρακτήρα που συμπεριλαμβάνονται στη στρατηγική για το 2020 απαιτεί πολύ συντονισμένες δράσεις και πρέπει να είμαστε πολύ στοχευμένοι στο πώ δαπανούμε τα διαθέσιμα κονδύλια. Διότι οι εδαφικέ και περιφερειακέ διαφορέ στην Ευρώπη είναι σοβαρέ. Για να καλυφθούν αυτέ οι διαφορέ, θα πρέπει να προσαρμόσουμε και εμεί λόγο στην αναπτυξική μα πολιτική. Αυτό λοιπόν το προφανές σχόλιο καθορίζει το πώς θα ολοκληρωθεί ο προσανατολισμός που θα λάβουμε. Ένας προσανατολισμός έχω τον, που τον βρίσκω λανθασμένο και επικίνδυνο. Δηλαδή, αδιακρίτως να πάρουμε τα κονδύλια και να τα υποβάλουμε όλα στους ίδιους κανόνες. Πίσω από αυτή τη δίκαιη αξίωση για συντονισμό μπορεί να υποκρύπτεται, και όντως υποκρύπτεται, η άποψη ότι Μπορεί να υπάρχει μια διάκριτη εδώ διαχείριση των κονδυλίων, κάτι το οποίο δεν συμμερίζομαι καθόλου. Τα κονδύλια λοιπόν του ΕΚΤ θα πρέπει να παραμείνουν ένα αυτό καθεαυτό εργαλείο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να έχει τους δικούς του πόρους και τους δικούς του κανόνες. Το να μετατραπεί σε ένα από τα πολλά ταμεία θα είναι ένα Ένα σφάλμα που μπορεί να μην βοηθήσει την πολιτική της απασχόλησης. Ή για να το πω πιο καλά, μπορεί να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα στην απασχόληση ποσοτικά. Αλλά εμάς δεν μας απασχολεί μόνο η αριθμητική αύξηση της απασχόλησης, αλλά και ποιοτική. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τον ανταγωνιστικό πρότυπο που θέλει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ποιότητα και του προϊόντος και των διαδικασιών και της εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πεπισμένος ότι όλα τα στοιχεία διάκρισης ακόμα και αυτά που μπορεί να οδηγήσουν σε γραφειοκρατικές καθυστερήσεις δικαιολογούνται, δικαιολογούνται λόγω του ιδιαίτερου μοναδικού χαρακτήρα που είχε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο από τη στιγμή τη ίδρυσή του. Βεβαίω, εάν χρησιμοποιείται λίγο το ταμείο αυτό, θα πρέπει να δώσουμε κάποια απόκριση. Αλλά η απόκριση δεν είναι να αλλάξουμε το χαρακτήρα του και τη φύση του, είναι να αλλάξουμε του μηχανισμού, του μηχανισμού ελέγχου. Θα έλεγα λοιπόν, ε, λόγω χάρη, ότι λογικό θα ήταν να πειραματιστούμε με λύσει που μπορεί να οδηγήσουν σε λιγότερους έλεγχους στην είσοδο, αλλά σε πολύ αυστηρές κυρώσεις, εάν αποδειχθεί τη στιγμή της επαλήθευσης, ότι έχει χρησιμοποιηθεί ένα κονδύλι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για λανθασμένους σκοπούς. Θα πρέπει λοιπόν να δίνουμε κονδύλια μεν, αλλά να τιμωρούμε εκείνους που στρεβλώνουν τον τελικό στόχο. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί εν ζωή αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ταμείου. Να μην ακούμε τις κολακίες και τις σιρήνες όσων φαντάζονται ότι με στοχευμένες δράσεις χρονικά και ποσοτικά καταλήξουμε να καταστρέψουμε εξαιτία όλων αυτών ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία που διαθέτουμε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στην κυρία Χάρκιν και την κυρία Λίν, την πρόεδρό μας. Ευχαριστώ. Έχω τέσσερις ερωτήσεις, αλλά μάλλον δύο από αυτές έχουν απαντηθεί. Για το ζήτημα της συμπληρωματικότητας με άλλα ταμεία να προσθέσω κάτι για το Ταμείο Μικροοικονομικών και τα, ταμεία, τα προγράμματα Τζέρεμι και Τζέσικα. Αυτά να ληφθούν υπόψη από την άποψη της συμπληρωματικότητα. Κάτι πρότεισε και ο κύριος Έρη για το τι είδου ε, στόχευση των δράσεων πρέπει να υπάρχει ώστε να μπορούν να καταμετρούνται τα αποτελέσματα. Τρίτο ερώτημα. Προς τον κύριο Γκάρσιν το δεύτερο ομιλητή μίλησε για το ΕΚΤ και είπε ότι δείχνει ένα νέο χαρακτήρα κοινωνικού και επαγγελματικού βίου στο πλαίσιο της πρόορης συνταξιδότησης. Εάν μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο σε αυτό. Και τελικό ερώτημα, και αυτό τέθηκε από όλους τους ομιλητέ, το ζήτημα του να έχουμε όσο περισσότερους συνομιλητέ ε, μπορούμε. Ε, Μίλησαμε για ένα φόρουμ για μη κυβερνητικέ οργανώσει, για τη στήριξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων, την τεχνική, να του δώσουμε δηλαδή ό,τι χρειάζονται. Και εγώ θα συμφωνούσα απόλυτα με κάτι τέτοιο. Επίση, ακούσαμε για την ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, ε, ευρωπαϊκό, εθνικό. Ταυτόχρονα, ακόμα για απλούστευση να γίνεται πολλή λόγο. Το δικό μου λοιπόν, δική μου ανησυχία είναι ότι όσο περισσότερο είναι συσχετισμοί, όσο περικρίκη τη αλυσίδα, τόσο περισσότερε δυσκολίε. Έχετε καμιά ιδέα για το πώ μπορούμε να πετύχουμε εξισορρόπηση μεταξύ των επιπλέον κρίκων της αλυσίδα και της ανάγκης για απλούστευση. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους ειδικού μας για τις παρουσιάσεις τους, διότι αυτή η συζήτηση είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Εδώ και καιρό συλλογιζόμαστε και σκεφτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνει εδώ παραλληλισμός, μάλλον να διαστούν οι ειδικοί των οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων. Από την άλλη όμως κάποιοι απέχουν από την αγορά εργασίας, έχουν παραμείνει για πολύ καιρό εκτός αγοράς εργασίας. Γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικέ μέθοδοι που να αξιοποιηθούν ώστε να προσεγγίσουν όλοι αυτοί πάλι την αγορά εργασίας. Την αγορά εργασίας. Τα συζητήσαμε όλα αυτά και είναι ένα καθοριστικό ερώτημα. Πώς πρέπει να δράσουμε για να έχουμε αποτέλεσμα. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία και να δούμε πώς χρειάζονται διαμεσολαβητές όπως οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ξέρουμε ότι οι περιφέρειες διαθέτουν πολλές κυβερνητικές, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που όμως πτώχευσαν γιατί χρησιμοποιούσαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και η υπερβολική γραφειοκρατία δεν τους επέτρεψε να ανθίσουν. Θα πρέπει να περιοριστεί λοιπόν και η γραφειοκρατία, να τονώσουμε την ευελιξία που είναι απολύτως αναγκαία. Συμφωνώ απολύτως και για την πρόληψη. Κάθε φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στηρίζει ένα πρόγραμμα, θα πρέπει εξ αρχής να προσφέρεται βοήθεια. Εάν η βοήθεια δίνεται καθυστερημένα, τότε δυστυχώς δεν ωφελεί συνήθως η κυρία Γκρίνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς ορισμένα ερωτήματα, γιατί κάποια ήδη τέθηκαν. Για το δημοσιονομικό χαρτοφυλάκιο. Προπολογισμό. Περισσότερα, τα ίδια, καλύτερη δαπάνη. Επίσης για τη χρήση του ΕΚΤ, η συγχρηματοδότηση σας φαίνεται να είναι ένας από τους τρόπους που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Επίσης, το Ταμείο αυτό θα μπορούσε να παρέχει βοήθεια ισότιμα σε όλα τα κράτη-μέλη, κάποιοι έχουν περισσότερα δικαιώματα λόγω μειωμένου ΑΕΠ. Και με το νέο κανονισμό που θα φτάσει στα μέσα του 2011 και τον το πεδίο δράσης του ΕΚΤ, ε, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει, θα πρέπει να είναι πιο δεσμευτικό και πιο συγκεκριμένο το πεδίο δράσης του ΕΚΤ. Διότι τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή μπορούν να συμπεριλάβουν ό,τι θέλουν λίγο πολύ. Και για τους δείκτες. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Ναι, να αλλάξουμε δείκτες, αλλά ποιους θα υιοθετήσουμε. Διότι όταν μιλάμε για την ποιότητα της ζωής, ε, πολύ δύσκολα καταμετράτε κάτι τέτοιο. Και είναι διαφορετικό από άνθρωπο σε άνθρωπο και από κάτω σε κράτο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, Ευχαριστούμε κυρία Γιαζοβλέσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό που ακούσαμε τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων, αλλά δεν μιλήσατε τόσο για τους δικαιούχους. Αναγνωρίζω ότι και τονίζω ότι αυτό είναι το σκέλος που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Ήθελα να ξέρω λοιπόν την άποψή σας σε σχέση με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής τις εκθέσεις μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει διαπιστώσει ότι το 70% των τελικών δικαιούχων είναι εργαζόμενοι με ενώτερε σπουδέ, ενώ μόνο 30% των δικαιούχων του Ταμείου είναι αυτοί που θα έπρεπε να προστατεύονται από το Ταμείο, οι άνεργοι δηλαδή, ω προ την πρόσβαση των ε, ανθρώπων με αναπηρίε στο ΕΚΤ. Ε, υπάρχουν πολλές διαφορετικές ε, δυνατότητε για αυτού του ανθρώπου που είναι μια πολύ ευάλωτη ομάδα και για άλλε ομάδε στόχου που είναι πιο δαπανηρέ. Ε, για του ανθρώπου αυτού χρειάζεται η δημιουργία ειδικών αιθουσών, ειδικέ υποδομέ, χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν να μην, παρά να συμφωνήσω με την ιδέα ότι το ΕΚΤ θα πρέπει να αφορά περισσότερο τις μη κυβερνητικές οργανώσεις Αλλά δεν θα συμφωνήσω με αυτό, διότι τα κονδύλια του ΕΚΤ πολλές φορές έχουν πλουτίσει κάποιες με κυβερνητικές οργανώσεις. Και μάλιστα σε... αφήνοντας εκτός ε, ωφελημάτων τους βασικούς δικαιούχους. Πρέπει λοιπόν να τονώσουμε το ρόλο του ΕΚΤ και να πάμε σε αυτή την σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ Πρόεδρε κυρία Ντελή. Ευχαριστώ και τους διάφορους ομιλητές για τις εξαιρετικές τους παρουσιάσεις. Εγώ θέλω να σταθώ στη συμπληρωματικότητα του ΕΚΤ και του ΦΕΝΤΕΡ, διότι είμαι μέλος και της Επιτροπής της ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Επιτροπή αυτή εξετάζει τώρα την δυνατότητα βελτίωση των κομιλίων του ΕΚΤ στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα ακριβώς να υπογραμμίσω την συμπληρωματικότητα του ΕΚΤ και του ΦΕΝΤΕΡ. Να δώσω το εξή παράδειγμα. Κοινοτικέ πρωτοβουλίε που έχουν ήδη αναλυφθεί. Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία Urban, η οποία είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συμπλήρωση των μέτρων του ΦΕΝΤΕΡ από τα μέτρα του ε, ΕΚΤ. Το πρόγραμμα Urban 1 και Urban 2 επέτρεψαν να υλοποιηθούν οι έννοιες της ε, κοινή προσέγγισης στα πλαίσια του προγράμματος αυτού. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια τέτοια κοινή προσέγγιση, ιδίω για τις ε, συνοικίες της μειονεκτούσας των πόλεων και προκειμένου να κινητοποιηθούν οι πολίτες και να είναι σε θέση να ανακαινήσουν ε, το πρόσωπο των συνοικιών αυτών, αλλά βελτιωθεί και η πρόσβαση στις υπηρεσίες και οι υποδομές. Όλα αυτά πρέπει να επαναργοποιηθούν. Πρέπει να επιμείνουμε εδώ στην διάσταση την αστική νομίζω. Είναι ένας δείκτης ο οποίος θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερος. Τώρα, βάσει αυτού του δείκτη, θα ε, καταπολεμήσουμε τις εδαφικές ανισότητες. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση κοινή, σφαιρική, η οποία να επιτρέπει ακριβώς σε όλους τους ε, παράγοντες, σε όλους τους συμμετέχοντες, σε όλους τους κατοίκους να έρθουν πιο κοντά. Να καλύπτονται οι ανάγκες τους και τα αιτήματά τους. Εδώ έχουμε μια θετικότατη αποτίμηση του προγράμματος αυτού, η οποία θα δημοσιευτεί τον 1η Δεκεμβρίου κιόλα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα στο οποίο θα μπορούσαμε να βασιστούμε χωρίς ε, ιδιαίτερε ανησυχίε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ έχω ένα-δυο ερωτήματα. Πώ νομίζετε ότι μικρέ μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπορούν να μάθουν για τα διαφορετικά προγράμματα, διότι αυτό είναι ένα τομέα που απασχολεί πολλούς ε, για συγκεκριμένε πρόοδου που μπορούν να αποτελεστούν. Η κυρία Σέτερ μίλησε για την ε, πρωτοβουλία Equal. Επίση, πώ μπορούμε να διευκολύνουμε την καλύτερη ανταλλαγή των πρακτικών, των καλών πρακτικών, εφόσον τόσα πολλά προγράμματα τρέχουν παράλληλα σε τόσο διαφορετικά κατημέλη. Ε, εδώ τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή γνώση για του ΜΑΕ και του ΔΕ. Θα σα δώσω και πάλι το λόγο και θα σα παρακαλέσω να περιοριστείτε σε δύο λεπτά ο καθένα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ε, αν υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να απαντήσετε, ίσω να μπορούσατε να μα στείλετε γραπτέ απαντήσει, αν δεν έχετε χρόνο τώρα. να στραφώ απευθείας στον κύριο Τορτουέρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες υποτυπώδεις απαντήσεις. Για το πρώτο ερώτημα, την ετήσια διάρκεια, πέντε χρόνια συν δύο, η θέση της Επιτροπής θα μπορούσε να είναι μια καλή λύση. Το δημοσιονομικό πλαίσιο φέτος μας φαίνεται εύστοχο για τα διαφορετικά μας προγράμματα. Το ΕΚΤ ανταποκρίνεται σε αυτό. Πέντε χρόνια φαίνονται λίγα. Πέντε συν πέντε με ενδελεχή, κατά λεπτομεριακή ε, αξιολόγηση στα μέσα της περίοδου είναι κάτι που φαίνεται λογικό. Σε ό,τι αφορά τη συμπληρωματικότητα του ΕΚΤ και του Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, η περίοδος ορίμανσης είναι πολύ μακρά. Θα πρέπει το ΕΚΤ να συμπληρωθεί, διότι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μπορούν να συμπληρωθούν. Συμπληρωματικότητα λοιπόν μεταξύ των διαφόρων επιδοτήσεων, πράγμα που θα μπορούσε να τονιστεί για να φανεί πώς ανταποκρίνονται οι δράσεις στην επίτευξη των στόχων. Εδώ όμω θέλουμε ένα εργαλείο συγκεκριμένο, ε, ταχύ, που απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων για το πρόγραμμα Equal και τις αρχές του. Βεβαίως, στην Ισπανία Ό,τι αφορά το ΕΚΤ, τα διαμετωμεακά στοιχεία, η ισότητα των ευκαιριών, ε, η λειτουργικότητα των ταμείων, όλα αυτά αφορούν το 2012 και 2013. Πρέπει να υπάρχει σαφής ε, κατάταξη των ε, προγραμμάτων του ΕΚΤ ανακατηγορία σε ό,τι αφορά την θετική διακριτική μεταχείριση υπέρ των γυναικών λόγου χάρη. τέτοιε δράσει εφαρμόζονται στην Ισπανία. Μια άλλη ερώτηση στην οποία θέλω να προσπαθήσω να απαντήσω είναι η διαχείριση της συμπληρωματικότητας των μικροοικονομικών και των δικτών θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι δείκτες να ορίζονται με τρόπο πολύ ακριβή σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε παρόμοιους ή και ταυτόσιμους δείκτες. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι συγκρίσιμοι οι δείκτες. Εάν το να επιτύχουμε τους στόχους μας υποχρώνει να πετύχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα πρέπει τότε οι στόχοι να είναι ήδη πολύ προσεκτικά διατυπωμένοι να είναι συγκεκριμένη. Το ΕΚΤ μπορεί να πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους πολίτες. Εάν αυτό έχει και οικονομικό αντίκτυπο, θα πρέπει να μην υπάρξει οποιαδήποτε απειλή από οικονομικές άποψεις για την Ευρώπη. Μια κοινή διαδικασία θα μπορούσε να επηρεάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Εάν λοιπόν θέλουμε αποτελέσματα για τους πολίτες, χωρίς να, φερέσουμε αφαιρέσουμε το στοιχείο του ελέγχου, θα πρέπει να πούμε ότι το ΕΚΤ είναι ήδη αποτελεσματικό, επιτρέπει την επίτευξη αποτελεσμάτων και εννοείται ότι θα είχα κι άλλα πολλά να συμπληρώσω, αλλά δυστυχώς λόγω του χρόνου που μου δόθηκε θα φροντίσω να σας απαντήσω γραπτός. Um, Ευχαριστώ. Έχουμε και του υπόλοιπου ομιλητέ τη μερική διαταξή Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο κύριος Γκαρσά. Πολύ γρήγορα να προσπαθήσω να θίξω πολλά από τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η κοινωνική πολιτική και η πολιτική της απασχόλησης είναι πάντοτε εθνικές. Το κοινωνικό ταμείο δίνει, πρικοδοτεί με μέσα τα διάφορα κράτη, βάσει συγκεκριμένων κανόνων. Αυτό σε επίπεδο κράτους αποκαθιστά την έννοια της συμπληρωματικότητας μεταξύ του κράτους του ίδιου στο ρόλο του και της ε, εξουσίας που έχει έναντι των περιφερειών, των επαρχιών, των νομών, των διαμερισμάτων, των ε, τοπικών οργανώσεων, όλων των δομών που υπάρχουν πάνω στην επικράτειά του. Αυτό μας οδηγεί σε μια προσέγγιση κοινή, ολοκληρωμένη. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι βρισκόμαστε πάντοτε όσο πιο κοντά γίνεται στον πληθυσμό. Αυτό λοιπόν το στοιχείο της ολοκληρωμένης προσέγγισης, της σφαιρικής προσέγγισης, όπου καλύπτονται όλα τα ψυχοκοινωνικά και εργασιακά προβλήματα, οδηγεί στο να μπορούμε να κοιτάξουμε και τα παιδιά και τι οικογένειε, τα προβλήματα τα επαγγελματικά, του ηλικιωμένου, τα προβλήματα κοινωνική ένταξη. Αυτή είναι η ενσωματωμένη προσέγγιση, κάτι που το συναντούμε και στον ΩΣΑ. Είναι ε, ε η σφαιρική αυτή επισκόπηση των προβλημάτων. Για να είναι η πολιτική μα σφαιρική και να μην τα πετάμε όλα σε ένα μεγάλο τσουβάλιο που θα χάσουμε τον μπούσουλα, θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένε μελέτε, συγκεκριμένε αναλύσει και να εισάγουμε έννοιε όπω η κοινωνική κερδοφορία εδώ θα επανέλθω στην έννοια αυτή. Η κοινωνική κερδοφορία θα πρέπει να βασιστεί σε μακροπρόθεσμα προγράμματα, δηλαδή να υπάρχουν στόχοι και δράσεις που να σχεδιάζονται με μακρινούς ορίζοντες. Αυτό νομίζω ότι απαντά και στο ερώτημα του κυρίου Νταρντά. Δηλαδή, αν έχουμε προγράμματα μακράς διάρκειας με στόχους σχετικά ακριβείς, μπορούμε να καταλήξουμε στην κοινωνική κερδοφορία με συγκεκριμένους στόχους προς πίτευξη. Επιδιωκόμενους στόχους, όχι από οικονομικής μόνον άποψη, αλλά στο επίπεδο των ανθρώπων. Ε, αυτή είναι η προσταθεμένη αξία που μπορούμε να συνεισφέρουμε στα άτομα ως προς την απασχόληση, την ποιότητα τη ζωής, ποιότητα ζωής η οποία προφανώς είναι υποκειμενική, όμως όταν μιλάμε για ποιότητα ζωής δεν μιλάμε μόνο για την υποκειμενική ποιότητα ζωής αλλά και για την ε, ποιότητα όπως την αντιλαμβάνεται το ίδιο το άτομο. Τώρα, πώς θα προσεγγίσουμε τον κόσμο της εργασίας με όσους έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας για διάφορους λόγους. Μέθοδος. Πολλές μέθοδοι υπάρχουν. Πρέπει να τις εντοπίσουμε. Μπορώ να τις ονομάσω, μπορώ να τις ονομάσουμε όπως θέλουμε, αλλά θα τις διακρίνουμε μεταξύ ενεργοποίησης, ε, επαναπροσαρμογής, ε, ένταξης και επαναδραστηριοποίησης και αυτό θα οδηγήσει στην συμμετοχή των ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Σε δύο λεπτά αυτά μπορούσα να σας δώσω στοιχεία απάντησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλος, ο κύριος Ντάντε. Και πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω λιγότερο από ένα λεπτό στη μου. Σε ένα μόνο πράγμα λοιπόν θα απαντήσω τη γραφειοκρατία, την ερώτηση για τη γραφειοκρατία, όπου θα πω ότι πρέπει να βρούμε το ορθό μέτρο, δηλαδή τον γραφειοκρατικό εκείνο μηχανισμό που είναι αναγκαίος και επαρκής ώστε να λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά δεν θα πρέπει βέβαια αυτό να επιβαρύνει εκείνους που καλούμεθα να στηρίξουμε. Αυτό θα ήταν λάθος. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με μία προστασία που θα τους παραχθεί. Έχουμε να κάνουμε ακόμα και με την ε, επιβάρυνση ακόμη περισσότερο αυτών των ανθρώπων. Δεν θα έχουν να κάνουν τη βοήθεια. βλέπουμε να υπάρχει μια πολλαπλή διαστρωμάτωση. ένα ακόμη οργανισμό έχει ε, ενταχθεί σε αυτή τη διαστρωμάτωση για τα δημοσιονομικά αρμόδια, αλλά αυτό το γεγονός ε, μπορεί βέβαια να εξασφαλίσει το ε, ελέγχου, αλλά επιβαρύνει ακόμη προς τι δομέ. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλους, την εξαίρετη παρουσίαση, λέει ο πρόεδρο. Ακούσατε και από τι ερωτήσει ότι θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πολλές ώρες ακόμη στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και τις ε, παρατηρήσεις σας. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι... Η νεολαία σε κίνηση ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευση και κατάρτιση. Κυρία Στάινρουκ, θέλετε το λόγο αμέσω, θέλετε να ακούσουμε τι ε, παρουσιάσει και μετά να κάνετε τι ερωτήσει σα. Τζον Μάρτιν πρώτα, εκ μέρου του ΩΣΑ. θα μας παρουσιάσει τις προτάσεις για την βελτίωση της απασχόλησης των νέων. Και μετά θα έχουμε την κυρία Σονέ, ε, η οποία θα κάνει την επόμενη ομιλία. Κύριε Μάρτιν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μεγάλη τιμή που μου κάνετε και εμένα και τη συναδέλφου που μας επιτρέπετε να είμαστε εδώ σήμερα μέσα Θα ήθελα να παρουσιάσω πρώτα κάποιες από τις μελέτες μας, από τα διδάγματα θα έλεγα, από τα όσα έχουμε κάνει στην αγορά εργασίας και πριν από την κρίση αλλά και μετά από τις 16 χώρες του ΩΣΑ. Παρακαλώ λοιπόν να περάσουμε στην πρώτη διαφάνεια. Και εδώ έχουμε 16 ε, χώρες του ΩΣΑ που καλύπτουμε, εκ των οποίων 9 είναι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακολουθούμε επίσης έναν ορισμό που έχει να κάνει με το πρώτο στάδιο ένταξης στην αγορά εργασίας με την ηλικία των 15 ή 16 ανάλογα με τη χώρα μέχρι των 16 ετών. Έχουμε 16 επιμέρους εκθέσεις, για την κάθε χώρα δηλαδή. Έχουν δημοσιευθεί όλες υπό το τίτλο ε, «Θέσεις εργασίας για τους νέους». Και για τον επόμενο μήνα προβλέπουμε την ολοκλήρωση ενός ε, ε, συνοπτικού, μάλλον συνθετικού τόμου ε, που θα καταγραφεί όλες αυτές τις μελέτες σαν έκθεση ε, και το τι επισημαίνουμε ως καλές πολιτικές επιλογές ή εσφαλμένες στον, στην προσπάθεια να βοηθήσουμε αυτούς τους νέους να μπουν στην αγορά εργασία. Μια πρώτη συνθετική παρουσίαση της έκθεσης αυτής παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στο φόρουμ υψηλού επίπεδου για τη χάραξη πολιτικής στις 20 Σεπτεμβρίου ε, στο Όστος επίπεδο Υπουργών και θα δείτε από την ε, ιστοσελίδα που αναφέρουμε στη σελίδα, στην διαφάνεια αυτή δώσει περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες για το όσο έχουμε πράξει. Στην επόμενη διαφάνεια ξεκινώ επισημένοντας μόνο κάποια πάγια τυποποιημένα δεδομένα ως προς την παρουσία της νεολαίας στην αγορά εργασίας. Το πρώτο πράγμα που θα έχει κανείς υπόψη, αλλά θα πρέπει να λησμονεί κιόλα δεδομένου του πόσο κατεπίγουσαν κατά σε αυτή τη στιγμή, ότι πριν από την κρίση είχαν σημειωθεί σημαντικές βελτιώσεις προς την παρουσία της αγοράς, στην αγορά εργασία των νέων σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ και είχαμε μειωτική τάση για την ανεργία των νέων πριν από την κρίση, σχεδόν σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Ταυτόχρονα όμως υπήρχαν και έμονα προβλήματα στην ενσωμάτωση αγοράς εργασίας κάποιων μεριδίων του πληθυσμού των νέων μας, ιδιαίτερα εκείνων που ε, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και έτσι εντοπίστηκαν, είχαν εντοπιστεί δύο συγκεκριμένες ομάδες νέων που αντιμετωπίζαν ιδιαίτερο, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο και δυσκολίες προς την ανταξίνα αγορά εργασίας. Είναι η πρώτη ομάδα αυτή που ονομάζουμε οι νέοι που ξέμειναν, έμειναν πίσω, και η δεύτερη είναι αυτή που παίρνει τον τίτλο ε, με κακή ενσωμάτωση», όχι ικανοποιητική ενσωμάτωση. Για να περάσω λοιπόν στην πρώτη ομάδα νέων, εκείνους που ξέμειναν, είναι οι νέοι οι οποίοι σορέυουν μια σειρά από μειονεκτήματα. Ασφαλώς ε, θα έχετε υπόψη σας τέτοια παραδείγματα στις χώρες σας. Είτε κάποιο παιδί που άφησε το σχολείο προώρα, είτε κάποιο παιδί που έρχεται από, ένα, από μια μειονότητα εθνοτική ή από ε, οικογένεια μεταναστών που ζει σε ε, μειονεκτικές περιοχές και που αντιμετωπίζει ψηλό κίνδυνο είτε να μην μπορέσει να μπει στην αγορά εργασίας είτε να μην μπορέσει να παραμείνει σε αυτήν. Ο δείκτης δε, ε, ο δείκτης καθρέφτης που χρησιμοποίησαμε ήταν η ομάδα NEETS, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν ούτε δραστηριότητα επαγγελματικοί, ούτε βρίσκονται σε διαδικασία κατάρτισης ή εκπαίδευσης και δεν έχουν ε, πτυχίο ή πιστοποιητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και έτσι εδώ η κύρια πολιτική επιλογή, την οποία εντοπίζουμε εμείς, είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να εξασφαλίσουν ένα αναγνωρισμένο πτυχίο ή δεξιότητα. Στην επόμενη διαφάνεια. Η ομάδα αυτή πριν από την κρίση αντιστοιχούσε στο 10% της ομάδας ε, νέων από 15 έως 29 ετών που είχαν σταματήσει τις σπουδέ τους. Και εδώ θα δείτε στον πίνακά μας ότι υπάρχει μια, κάποια διαβάθμιση μεταξύ των κρατών που εξετάσαμε ως προς το μέγεθος της εν λόγω ομάδας και θα περάσω τώρα στη δεύτερη ε, ομάδα που είναι οι νεήλιδες με περιορισμένη ενσωμάτωση, με κακή ενσωμάτωση. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με νέους που έχουν συνήθως ε, πτυχίο δευτεροβάθμιας ενώτερης εκπαίδευσης και όμως ακόμη και σε περιόδους υψηλής ε, οικονομικής ανάπτυξης δεν μπορούν να διατηρήσουν παρά μόνο προσωρινές θέσεις εργασίας με δίκτυ καθρέφτη, όπως τον ονομάζουμε πρόξενη Indicator, 8% των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15-29 ετών πριν ακριβώς από την κρίση το 2005 με 2007, είχαν εγκαταλείψει τις σπουδέ τους και ε, εργάζονταν σε μια προσωρινή θέση εργασίας και που δύο χρόνια αργότερα δεν είχαν βρει μόνιμη δουλειά. Δηλαδή ένας νέος είχε αφήσει τις σπουδέ του, είχε πάρει μια προσωρινή σύμβαση, σύμβαση ορισμένου χρόνου και δύο χρόνια μετά ήταν ακόμα σε σύμβαση ορισμένου χρόνου ή ήταν άνεργος πλέον. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το μέγεθος αυτής της ομάδας σε ορισμένες χώρες όπου υπάρχουν πολλά εμπόδια ως προς τους ε, νεήλιδες, δηλαδή δεν είναι εύκολο κάποιος που δεν βρίσκεται στην αγορά εργασίας να βρει μια θέση, ε, έχουμε πολύ πιο έντονο το φαινόμενο αυτό και πιο μεγάλη την ομάδα όπως στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία. Και εδώ ε, εντοπίζουμε ακριβώ τον τρόπο με τον οποίο, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασία στο πρόβλημα. Δηλαδή είτε κλείνει την πόρτα είτε περιορίζει την πρόσβαση στου ανθρώπου αυτού. Άρα θα πρέπει η αγορά εργασία να αλλάξει, ο τρόπο λειτουργία τη αγορά εργασία. Στην επόμενη διαφάνεια, πριν ακριβώ από την κρίση, 8% των νέων τη Ευρώπη, όπω σα είπα νωρίτερα, ανήκαν σε αυτή την ομάδα ε, ηλικία και δεν είχαν ε, την δυνατότητα να μπουν σε μια θέση εργασία ε, τουλάχιστον μόνιμη. Στη δε επόμενη διαφάνεια θα δείτε ότι ένας εκ των πέντε νέων ανήκε σε μία από τις δύο ομάδες που προανέφερα. Δηλαδή είχαν εγκαταλείψει τις σπουδέ τους και αντιμετώπισαν σοβαρό κίνδυνο ε, δυσκολιών στην αγορά εργασίας. Και έτσι είναι βέβαιο ότι με την κρίση οι ομάδες αυτές έχουν αυξηθεί έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Ε, εκτιμήσεις μόνο μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ως προς το μέγεθος ε, την έκταση των ομάδων αυτών. Πάντως, ένας στους τέσσερις ε, νέους σήμερα φαίνεται ότι εντάσσεται σε, αυτή τη, αυτές τις δύο ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ονομάζουμε. Ας περάσω τώρα στην ε, στις επιπτώσεις των αντίκτυπο της κρίσης με την επόμενη διαφάνεια όπου νομίζω ότι δεν χρειάζεται εγώ να αναφέρω πως η παγκόσμια κρίση έχει πλήξει βαρύτατα τους νέους και τις προοπτικές τους για απασχόληση και ότι το μέλλον φαίνεται μάλλον ζωφερό. Η τελευταία μας εκτίμη προβολή δείχνει ότι για τους προσεχείς τουλάχιστον 18 μήνες θα παραμένει υψηλή η ανεργία των νέων που ήταν μάλλον με τρίων διαστάσεων μέχρι τώρα και με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεργία των νέων που ανήκουν σε αυτές τις δύο ομάδες. Και εδώ έχουμε να εξετάσουμε την ε, μακροπρόθεσμη επίπτωση, το μακροπρόθεσμο, το μακροπρόθεσμο τραύμα όπως ονομάζεται, δηλαδή την περίπτωση ε, κάποιος άνθρωπος ο οποίος έστω και όταν έχει τελειώσει η κρίση να μην μπορεί να ξεφύγει από τα προβλήματα τα, τη δυσκολία στο να βρει μια θέση εργασίας ή μια θέση εργασίας με ικανοποιητικές αποδοχές και ότι αυτές οι αποδοχές του θα είναι πάντοτε χαμηλότερες από τους άλλους νέους που είχαν καλύτερη, καλύτερες ευκαιρίες και τύχη. Προχωρώ για να σας αναφέρω τις τελευταίες μας προβολές που δείχνουν ότι τα ποσοστά ανεργίας στους νέους μπορεί να φτάσουν του χρόνου στο 23% και δεν προβλέπεται να μειωθεί αυτό το ποσοστό ανεργίας πριν από τις αρχές του 2012, ίσως και τα τέλη του 2012 με αυτές τελευταίες μας προβολές και εκτιμήσεις. Τώρα, τι σημαίνει αυτό ως προς τις κύριες και βραχυπρόθεσμες προκλήσεις πρώτη προτεραιότητα που εντοπίζουμε με το έργο μας και που επαναλαμβάνουν και οι υπουργοί μας στο Όσλο λέει πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου από τα παιδιά, δηλαδή να μην δημιουργήσουμε, να μην επιτρέψουμε να δημιουργηθεί αυτή η τραυματισμένη γενεά. Δεύτερον, κάποιοι νέοι αποφασίζουν να αντιδράσουν στην κρίση μένοντας για πιο μεγάλο διάστημα στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια ε, επένδυση καλή μεν, που όμως θα πρέπει να φροντίσουμε να τους προσφέρει τις δεξιότητες και την εμπειρία που θα είναι όντως χρήσιμη όταν μπορούμε, να πούμε ότι έχει εξασφαλιστεί μια κάποια, ένας κάποιος καλός ρυθμός ανάκαμψης. Τρίτον, τα μέτρα για την αργορά εργασία και ιδιαίτερα αυτά τα οποία είναι εστιασμένα στους ε, νέους προς αυτή τη δυσκολία θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά και να διατηρήσουν ε, μία στάση ενεργοπιδραστηριοποίηση, δηλαδή να επιτρέπουν στους νέους αυτούς να μπουν πράγματι στην αγορά εργασίας και να αναλάβουν ε, θέσεις Και επίσης εν τέλει να εξασφαλιστεί ένα δίκτυο ασφαλείας με την, ε, και στην απασχόληση αλλά και στην κατάρτιση για τους νέους που μένουν άνεργοι ή που μόλις έχουν μπει στην αγορά εργασίας τι θα πρέπει να κάνουν οι χώρε για να επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Καταρχάς πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία να προχωρήσουμε με μια ταχεία και επιλεκτική ε, παρέμβαση ώστε να βοηθήσουμε αυτού του νέου να παραμείνουν σε επαφή με την αγορά εργασίας. Ε, είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι νέοι και μάλιστα να του εντοπίσουμε εγκαίρω και να εντοπίσουμε εγκαίρω ποια είναι η πιο αποτελεσματική παρέμβαση. Να του προσφέρουμε αρρωγή στην αναζήτηση θέσεις να παρατείνουμε την προσωρινή ε, προστασία από την ανεργία και τα, και, και τα προβλήματα τα κοινωνικά για εκείνους τους νέους οι οποίοι δεν έχουν επαρκή προσόντα ή έχουν εξαντλήσει το, την περίοδο υποστήριξης και να βοηθήσουμε κυρίως τους μαθητευόμενους που έχουν απολυθεί, που επιτοπλίστων ε, εντοπίζονται στον χώρο τον κατασκευαστικό και τον οικοδομικό, που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση, και ως εκ να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τις ε, δεξιότητές τους. Εν τέλει δε, απαραίτητο είναι να συζεύξουμε σε ευχθή το δυναμικό αυτό ε, με το δίκτυο ασφαλείας, με αυτό που ονομάζουμε στον ΩΣΑ μία προσέγγιση αυστηρή προσέγγιση αμοιβαίων υποχρεώσεων, δηλαδή ένας νέος ο οποίος έχει φοληθεί από μια τέτοια κοινωνική στήριξη και προσέγγιση να μπορεί να ε, βρει μόνο στις εργασίες να βελτιώσει τις ε, δεξιότητες και την αποσχολησιμότητά του. Στην επόμενη διαφάνεια, προχωρώντας στο μέλλον και όταν ε, αρχίσει να βελτιώνει τους ρυθμούς της η είπε να την ικανοποιητική ρυθμή ανάπτυξη, θα δούμε μια σειρά από προβλήματα που θα, κληθούν, ε, κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη και άλλες χώρες του ΩΣΑ. Με πρώτο, ζωτική σημασία στο να βεβαιωθούμε ότι κάθε ένας που θα φεύγει από την, ε, από την ε, εκπαιδευτική διαδικασία, το εκπαιδευτικό σύστημα, θα έχει επαρκείς δεξιότητες για την αγορά εργασίας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να υπολογίσουμε αυτό το πράγμα και να εξασφαλίσουμε τις επαρκείς δεξιότητες, ε, αυξάνοντας το, την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 16, 18 ή 19 χρόνια. Αυτό, κατά την άποψη του μπορεί να είναι χρήσιμο μέσο για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, εφόσον όμως, εφόσον όμως είναι συνδεδεμένος με την απόκτηση δεξιοτήτων για τον εν λόγω νέων. Να μένει δηλαδή ο νέος περισσότερο διάστημα στην διαδικασία της εκπαίδευση ή της κατάρτιση, αλλά μόνο με προϋπόθεση ότι αποκτά νέε δεξιότητες, επιπλέον και επαρκείς δεξιότητες. Δεν θα τον υποχρεώνουμε το νέο με το ζόρι να κάθε μια ώρα παραπάνω μέσα στην ε, τάξη του σχολείου, ειδικά εάν έχει για κάποιους λόγους ε, δυσκολευτεί στην ε, μαθητιακή του πορεία. Και έτσι προωθούμε την ευκαιρία για μια, μια, μια δεύτερη ευκαιρία για εκπαίδευση και κατάρτιση για παιδιά με περιορισμένες δεξιότητες, για νέους μετανάστες και δίνουμε μερικές φορές μια δεύτερη ευκαιρία έτσι ώστε να βοηθήσουμε ότι να βοηθήσουμε ώστε ε, φεύγοντας από το σχολείο το παιδί, από το εκπαιδευτικό σύστημα να έχει σημαντικές αξιόλογες δηλαδή δεξιότητες. Ένα άλλο πράγμα που θα πρέπει ιδιαίτερα να μας απασχολήσει είναι η μετάβαση από το σχολείο στο χώρο εργασίας να είναι λιγότερο απότομη. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερε ευκαιρίες για τον νέο. Θα μπορεί ο νέος να συνδυάζει περισσότερο την ε, απασχόληση με την μάθηση, με την εκπαίδευση. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που λένε ότι ο συνδυασμός με κάποια, κάποια υπογραμμίζω δουλειά ε, των σπουδών έχει χρησιμότητα, εφόσον βέβαια ο, η επιβάρυνση στη μελέτη του παιδιού δεν είναι υπερβολική. Φερρυπίν ε, γίνεται λόγος για ένα όριο των 15 με 20 το πολύ ωρών που, εργασίας του νέου που δείχνει ότι ε, μπορεί να τον ε, βοηθήσει στις σπουδέ του και ως προς την εμπειρία που θα έχει αποκτήσει αλλά και ως προς το ε, ποσό που θα μπορέσει να συλλέξει από την αμοιβή του και που θα τον βοηθήσει περισσότερο. Και αρκετοί θα είναι οι νέοι οι οποίοι θα μπορούν να συνδυάσουν την, τις σπουδέ με την εργασία. Και έτσι θα έχουμε μια πιο απρόσκοπτη μετάβαση στο χώρο εργασίας. Στην επόμενη διαφάνεια είναι πολύ σημαντικό πιστεύω η φραγμή ως προς τη ζήτηση θέσης εργασίας που αντιμετωπίζουν οι νέοι και που τους εμποδίζουν από την πρόσβαση ή από τις πραγματικές προοπτικές μιας σταδοδρομίας να αντιμετωπιστούν. Φέρει πίν. Υπάρχουν διακρίσεις που επιβάλλονται προς την πρόσληψη νέων, ιδιαίτερα ε, νέων με διαφορετική εθνοτική προέλευση, μειονοτική δηλαδή, ή μετανάστες. Είναι απαραίτητο αυτό. Επίσης είναι απαραίτητο να μειωθεί το κόστος απασχόλησης ε, νέων με χαμηλά πρόσοδα και χαμηλή παραγωγικότητα και αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους ε, τρόπους, είτε με την εισαγωγή, την επέκταση ε, μισθών κατώτερων από τον κατώτατο ή και χαμηλότερων κοινωνικών δαπανών, εισφορών δηλαδή, για αντίστοιχου μισθούς. Και επίσης, συμπληρωματικά ή υπαλλακτικά, να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αναζήτηση διαδικότητας, δηλαδή ταυτόχρονες λειτουργίες και παρουσία στην αγορά και την, ε, ε, μεταξύ αγοράς και εργασίας. Έχουμε πολλά λοιπόν να κερδίσουμε από καλά συστήματα κατάρτισης, μαθητείας δηλαδή των νέων, που ήδη βλέπουμε σε αρκετά τα οποία επενδύουν και προσπαθούν να τα καταστήσουν, να τα διατηρήσουν ως αποτελεσματικά μέσα για τον νέο, για τη μάθηση. Όμως πέραν αυτής της περίοδου της μαθητείας πρέπει να εξασφαλιστεί πέραν μάλλον τη περίοδου αυτή τη κρίση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα είναι διατεθειμένε οι επιχειρήσει να προσφέρουν μαθητεία για του νέου και ότι θα επιλέγουν για τη μαθητεία αυτή και παιδιά από μειονοτικέ οικογένειε ή από ε, το χώρο των μεταναστών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πολλαπλό μέρισμα όπως ονομάζουμε γιατί και ο εργοδότης κερδίζει και βελτιώνει την, ε, το κόστος και την αποτελεσματικότητά του και δίνει την ευκαιρία για κατάρτιση και μαθητεία σε ένα νέο στον οποίο επενδύει και ο οποίος νέος μπορεί να είναι μερικές φορές και τυχερός εφόσον είναι ο εργοδότης του διατεθειμένος να τον κρατήσει στην ίδια θέση όταν ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος μαθητείας ή και από την άλλη εφόσον ακόμη φύγει ο νέος μαθητευόμενος έχει ήδη ε, αποτελέσει αυτή η μαθητεία εφαλτήριο για μια καλύτερη θέση εργασίας. Και βέβαια υπάρχει και μια κάποια οικονομική ε, ωφέλεια με την έννοια ενός μισθού, μιας αποζημίωσης, ενός χαρτζηλικιού που δίνεται στον μαθητευόμενο. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχει τεράστια σημασία, ζωτική σημασία το να επενδύσουμε στην ε, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητευόμενους ε, και αντίστοιχα τέτοια προγράμματα. Και για να ολοκληρώνω, Πρόεδρε, με τελική μου διαφάνεια, θα ήθελα να επισημάνω τέσσερις παρατηρήσεις. Όντως, ε, οι περισσότερες χώρες του ΑΣΕ, του ΩΣΑ, <coughs> αντιδρούν στην κρίση ενισχύοντας τους πόρους για τα προγράμματα που απευθύνονται στην νεολαία. Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό αυτή η ορμή που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή, αυτή, αυτό το ενδιαφέρον, να μην εγκαταληφθεί. Και είναι ακόμη πιο κατεπίγουσα η ανάγκη ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που χωρών, ε, χωρών ε, οι οποίες έχουν την ανάγκη να περικόψουν ε, το δημόσιο του έλλειμμα, να μειώσουν το εξωτερικό τους χρέος και έτσι τέτοιου είδους πόροι που αφιερώνονται στους νέους θα πρέπει να διατίθενται κατά τρόπον αποτελεσματικό. Τρίτο τομέα τρίτη παρατήρηση, είναι σημαντικό πιστεύουμε να γίνονται επενδύσεις στην πρόληψη ώστε τα περισσότερα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο να μην μπαίνουν στον κικαιώνα της ε, αδράνειας ή της ανεργίας. Ο στόχος όμως, ε, η ομάδα όμως στόχος για εντατική στήριξη θα πρέπει να είναι η κύρια αυτή ομάδα νέων, στους οποίους βλέπουμε σωρευτικά κάποια μειονεκτήματα και ιδιαίτερα να ε, έχει σημασία να περιγραφεί ο τύπος αυτού του νέου που βρίσκεται στην πιο δύσκολη κατάσταση και να εντοπιστεί ώστε να προσφερθεί η διαχείριση των περιπτώσεων αυτών, η περιγραφή τους, η στήριξή τους και η ενθάρρυνση που χρειάζονται για να μπουν στην αγορά εργασία. Κυρία Πρόεδρε, κλείνω έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ και σημειώνω ότι με πολύ μεγάλη χαρά να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε να μας υποβάλλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Τάνεκ. Να πω ότι έχουν έρθει έξι φοιτητές από την περιφέρειά μου. Του Ράκμπι. Vielen Dank, ähm, äh, κυρία Στάνζουκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ ως ε, συντάκτη αυτής της νομοδότησης. Ε, ε, έχω αρχίσει από τον Απρίλιο ήδη να μελετώ την έκθεση του Οσάκη. σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ήταν πολύ χρήσιμη και μας προσφέρει πολύ σημαντικό υλικό για τη συζήτησή μας. Έχουμε, εκατοντάδες εκατομμύρια, έχουμε εκατομμύρια νέους στην Ευρώπη, 20% εκ των οποίων είναι άνεργοι αυτή τη στιγμή και οι επιπτώσεις αυτή τη ανεργία δεν αφορά μόνο τον, τον την οικογένειά του, αλλά και το ίδιο το κράτος μέλος. Ήδη στην έκθεση σα το αναφέρατε, Πολλοί από τους νέους αυτούς δεν έχουν, αφού αφήνουν το σχολείο ή ολοκληρώσουν τις σπουδέ τους, καν την ευκαιρία να ξεκινήσουν ε, με μια θέση εργασίας, να μπουν στην αγορά εργασίας και έτσι μπορούμε να μιλήσουμε για ορισμένους από αυτούς για ε, μια χαμένη γενιά. Γι' αυτό καλό θα είναι να βρούμε τα μέσα να αποτρέψουμε τέτοιου είδους φαινόμενα εγκαίρως. Επίσης, ε, η έναρξη σταδιοδρομίας για τους νέους αυτούς ξεκινά, σημαίνει πολλές φορές θέσεις εργασίας ε, ε, επίφοβες, θέσεις εργασίας όχι ασφαλείς. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν την προσπάθειά μας, έχουμε μελετήσει με επίκεντρο τους ε, νέους και μπορούμε χάρη στα δικά σας και στις προτάσεις να έχουμε περαιτέρω συζήτηση. Έχει περάσει η ώρα όμως mm. και ξέρω ότι θα συζητήσουμε διεξοδικά και άλλα θέματα Γι' αυτό θα περιοριστώ σε τρία ερωτήματα προς εσάς. Όπως λέει η έκθεσή σας, το 2010-2011 θα είναι τα δύο ε, έτη στα οποία θα σημειωθεί η υψηλότερη ενεργεία των νέων. Η κατάσταση για διάφορους λόγους ε, και λόγω της ε, διεξόδου από την κρίση που προβλέπατε αλλά και λόγω των δημοκρατικών εξελίξεων θα ανατραπεί μετά το 2011. Θα προλάβουν όμως αυτά τα παιδιά να πιάσουν το τρένο της ζωής. Και δεύτερη ερώτηση, μιλήσατε για κίνητρα για τον εργοδότη, έτσι ώστε να τον ενθαρρύνουμε μέσω φορολογικών απαλλαγών, μείωση του, του εργασιακού κόστους κτλ. να προσλαμβάνουν περισσότερους νέους. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς την απασχόληση των πιο ηλικιωμένων το να βοηθήσουμε τους νεότερους καλό θα ήταν να μην οδηγήσει σε μια σύγκρουση μεταξύ των γενεών. Και τελευταία ερώτηση. Από την ε, μελέτη, από την έρευνα του ΟΣΑ, φαίνεται ότι υπάρχουν χώρες ε, οι οποίες είναι σε θέση καλύτερα να διαχειριστούν την ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων. Μπορούν καλύτερα να τους στηρίξουν στην προσπάθεια αυτή μπορείτε να μας εντοπίσετε αυτά τα κράτη και βέβαια εγώ έχω σημειώσει ε, τη δική μου την πατρίδα τη Γερμανία όπου πιστεύω ότι έχουμε καλύτερες επιδόσεις χάρη στο διαδικό λεγόμενο σύστημα που συνδυάζει θεωρητικές σπουδές, σπουδές αλλά και για μαθητεία στους ε, νέους μας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Τέρνεν και μετά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα μελέτη από τον ΩΣΑ, μια παρουσίαση η οποία ασφαλώ μπορεί να δώσει αρκετές απαντήσεις στο πλαίσιο και τα Μερικές φορές τραγικά δεδομένα τα οποία βλέπουμε, δόθηκε μια περιγραφή ήδη. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον αυτή η κρίση που αντιμετωπίσουν οι νέοι και στον τομέα της απασχόλησης θα περιοριστεί στα δύο έτη, το 2010-2011 και κατά πόσον θα είναι να ξεφύγουν από αυτή αμέσω μετά. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε μακροπρόθεσμα φαινόμενα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται παρά μόνο αν προσφερθούν επαρκείς δυνατότητες κατάρτισης και ε, συμπληρωματικής εκπαίδευσης μεσοπρόθεσμα δηλαδή, μάλλον βράχη πρόθεσμα δεν βλέπω να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Εδώ θα ήθελα εγώ να αναφερθώ περισσότερο στην τρίτη ομάδα, δηλαδή εκείνη η οποία έχει την κατάρτιση και όμως δυσκολεύεται να βρει θέση εργασίας. Παρότι ξέρουμε ότι σε ορισμένου τομεί λείπουν εξειδικευμένα ε, εργατικά χέρια ή εργατικό δυναμικό. Ίσως εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερο με το πρόβλημα της λειτουργίας της αγορά εργασίας, της διαχείρισης αγοράς εργασίας και του προσανατολισμού των σπουδών στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ένα ερώτημα και επίσης είπε ο κύριος Μάρτιν ότι τα κράτη-μέλη δεν περικόπτουν τα κονδύλια που διαθέτουν για την εκπαίδευση των νέων. Όμως εγώ έχω υπόψη ορισμένε περιπτώσεις κρατών μελών τα οποία λόγω ακριβώς των δημοσιονομικών τους δυσκολιών προβαίνουν σε περικοπές των σχετικών ε, προγραμμάτων. Και το ίδιο βλέπουμε και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε. κυρία Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για την έκθεση για την νεολαία που εγκρίναμε τον Ιούλιο στο Κοινοβούλιο και ασχολήθηκα με πολλά από τα ζητήματα που θίξατε κι εσείς. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση στην Επιτροπή μας και έχω αρχίσει να απογοητεύομαι γιατί πραγματικά από πολιτικής, απόψεως, από απόψεως είναι κατεπήγον παρά το γεγονός ότι έχουμε οικονομικούς περιορισμούς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως ε, είναι να ε, επιμείνουμε και να δείξουμε την ευρωπαϊκή μας προστιθέμενη αξία και αυτό έχει να κάνει και με την ταχύτητα εφαρμογής, αλλά πρέπει να δούμε και τι είδους ε, πρωτοβουλίες πρέπει να τύχουν χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το να μπορέσουμε λοιπόν να διατηρήσουμε αυτή την ε, νεολαία σε για την οποία μιλούμε, ειδικότερα σε θέματα απασχόλησης, είναι ε, πραγματικά κατεπήγον ζήτημα για μένα. Και θα ήθελα να περάσω τώρα σε μερικά σχόλια επί της παρουσίασης και επί των προκλήσεων που αναφέρονται. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε, αλλά έχω και μερικές ερωτήσεις σχόλια. Στη σελίδα 11 που λέτε ότι πρέπει να προετοιμάσουμε τους Ευρωπαίους νέους για να είναι ε, έτοιμοι για να αναλάβουν θέσεις, ε, να λάβουν, θέσεις απασχόλησης όταν θα αρχίσει η ανάκαμψη από την ε, οικονομική κρίση γιατί λέτε ότι υπάρχει περίπτωση να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν για απασχόληση. Κοιτάξτε, Μα τα κράτη-μέλη κόβουν, κάνουν περικοπές στον προπολογισμό από την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι ισχύει για όλε τι χώρε ευρωπαϊκέ, ε, όλε τι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τουλάχιστον σε πέντε χώρε που γνωρίζω ισχύει αυτό που λέω. Και είναι γεγονό ότι η εκπαίδευση είναι κάτι που πρέπει να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση. Άλλωστε εμείς δεν ε, είμαστε υπέρ της χαμηλόμης της εργασίας. Εμείς προάγουμε και ε, υψηλών προδιαγραφών θέσεις απασχόλησης και υψηλόμισθες. Πρέπει να είμαστε επίση πιο αποτελεσματικοί και από, απόψε ω κόστου. Γνωρίζω ότι σε πολλά κράτη-μέλη, εδώ και πολλά χρόνια, το βασικό πρόβλημα είναι όπως έχει αποδειχθεί από πολλούς ερευνητές, ότι αυτά τα μέτρα, τα πάρα πολύ δαπανηρά ε, για την αγορά εργασίας δεν λειτουργούν στην πράξη. Και αυτό το διαπιστώσαμε προσφάτως στην ε, Δανία. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν τι λειτουργεί κάθε φορά. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή απλώς να ξοδεύουμε χρήματα χωρίς να έχουν κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει να ξέρουμε, ε, να έχουμε υπόψη μας και τη διάσταση της ποιότητας όταν μιλάμε για πολιτικές, για ε, αποτελεσματικές πολιτικές για την αγορά εργασίας. Ένα ακόμη σχόλιο έχω για τη σελίδα 14, για την μείωση του ε, ε, και, ε, της, και των κοινωνικών εισφορών των πιο χαμηλόμισθων εργαζομένων. Κοιτάξτε, εδώ διαφωνώ καθέτο στο να υπάρχει μία δεύτερης κατηγορίας αγορά εργασίας για τους μετανάστες ή για τους νέους. Δεν είναι μία λύση, είναι κοινωνικός αποκλεισμός. Δεν αποδέχομαι αυτή τη λύση και θα ήθελα να μου εξηγήσετε ε, μου πείτε τη γνώμη σας για τους κινδύνους ε, μιας τέτοιας λύσης, γιατί για μένα δεν αποτελεί λύση από πολιτικές απόψεις. Μπορεί οι εργοδότες να το βρουν πολύ ελκυστικό ως λύση, αλλά εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε να υπάρχει μια δεύτερης κατηγορίας αγορά εργασίας για μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ως και οδησηγήτρια ως εισηγήτρια για την επαγγελματική κατάρτιση και την ε, μετεκπαίδευση ήμουν την περασμένη εβδομάδα μια αντιπροσωπεία στη Θεσσαλονίκη Σεντεφόπ, όπου βέβαια συζητήθηκε το θέμα αυτό της ενεργείας των νέων. Και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τη συνάδελφο. Η κατάσταση πραγματικά μας ε, γεννά μόνο απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Βλέπουμε ότι ε, ένα πρόβλημα το οποίο προϋπήρχε με την κρίση τώρα απλώς οξύνεται, επιδεινώνεται και λίγο πολύ οφείλεται σε μια σειρά από εσφαλμένες ε, πολιτικές επιλογές και πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη διαπιστώνουν ήδη σοβαρή ε, ανεργία των νέων. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα περιοριστεί μόνο στα λίγα πρώτα κράτη που, όπου φαίνεται τώρα υψηλό επίπεδο ανεργίας, αλλά θα επεκταθεί παντού και θα έχουμε σε λίγα χρόνια ανθρώπους που θα είναι 30 ετών και άνω και δεν θα έχουν μπορέσει καν να ξεκινήσουν μια σταδιοδρομία, να μπουν στην αγορά εργασία. Τι θα την κάνουμε αυτή τη γενιά, πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη γενιά που δεν θα εξαφανιστεί, απλώ θα συνεχίσει να ζει στα επόμενα χρόνια. Και το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι υπάρχουν καλά σχέδια πολλά καλά σχέδια που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας, τα παιδιά εκείνα που έχουν αφήσει το σχολείο, τα οποία ενδεχομένως δεν μπορούσαν να ενταχθούν καλά στο εκπαιδευτικό σύστημα, να τους δώσουν ένα τρόπο ε, να εξασφαλίσουν νέες δεξιότητες, επιπλέον προσόντα, και μάλιστα και κατά τρόπο που και το σχολείο μπορεί να επωφεληθεί εάν βοηθήσει το παιδί αυτό να μείνει στην εκπαίδευση και να με τη διακόψει μπορεί να έχει ένα σχολείο την δυνατότητα να βρει εφάνταστες λύσεις, εφόσον δει ότι έχει και το ίδιο συμφέρον και έτσι να βοηθήσει να μείνει ένα την στην εκπαίδευση. Εδώ λοιπόν μπορούμε να αναπτύξουμε δράσεις και σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να υποχρώσουμε κανέναν φυσικά να προσλάβει νέου ε, εργαζομένου, αλλά μπορούμε να, να πείσουμε τους εργοδότες ότι έχουν και κοινωνική ευθύνη και πρέπει να συμβάλλουν με την ε, επιλογή νέων εργαζομένων. Επίσης κάτι που είδα στην αντιπροσωπεία και στην αποστολή αυτή είναι ότι πολλά πράγματα γίνονται σε επίπεδο ε, τοπικό εφόσον συνεργαστούν όλοι οι παράγοντε κατά τρόπο συντονισμένο, δηλαδή και το σχολείο, μάλλον και ο παιδικό σταθμό για το σχολείο και ο εργοδότη. Ε, όλοι αυτοί οι παράγοντε πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συντονιστούν στις προσπάθειές τους και εδώ μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, να προσφέρει και να δώσει την έμφαση. Βεβαίως έχουμε ήδη τη λειτουργία και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην υπόθεση αυτή, αλλά έχουμε και άλλα πιλωτικά προγράμματα τα οποία μπορούμε για την προσεχή περίοδο να προγραμματίσουμε και να πούμε ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουμε τις ευκαιρίες δικτύωσης ε, των νέων, δικτύωσης των συστημάτων ενίσχυσης των νέων Γιατί αυτό είναι που ε, λείπει. Καλά προγράμματα υπάρχουν. Μερικές φορές δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια. Και εμείς ως Κοινοβούλιο, εάν θέλουμε να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα, θα πρέπει να δώσουμε αυτή την επιπλέον ε, προσθέμενη αξία. Και όχι απλώς να περιοριστούμε στο να συστήσουμε το θέμα για πέμπτη ή έκτη φορά εδώ. Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Εγώ έχω πολλές παρατηρήσεις. Καταρχάς, η φτώχεια των νέων. Είναι σωστό ότι πρέπει να πολεμήσουμε ώστε οι νέοι να έχουν δουλειά. Όμως αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα δυστυχώς ακόμη και όσοι δουλεύουν, όσοι εργάζονται, έχουν επισφαλείς θέσεις εργασίας και αμείβονται πάρα πολύ άσχημα. Άρα το ποσοστό φτώχειας είναι τόσο σημαντικό που θα πρέπει να βρούμε μέτρα συγκεκριμένα βελτίωση της ζωής των νέων αυτών. Δεν έχουν πρόσβαση καν σε υγειονομική περίθαλψη. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Είναι λοιπόν περίεργο να ξεκινάμε συζήτηση για επιδότηση αυτονομίας και εισόδημα αυτονομίας, συγγνώμη, γιατί εννοείται ότι οι νέοι πρέπει να είναι αυτόνομοι. Για να επανέλθω στην εκπαίδευση. Το είπατε, διανύουμε περίοδο κρίσης. Θέλουμε να μειώσουμε το δημόσιο έλλειμμα. Δεν επενδύουμε πια στην νεολαία. Και έχουμε καιρό να επενδύσουμε στην εκπαίδευση. Θα επανέλθω σε κάτι που κι εσείς είπατε. Είπατε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ανακτήσουμε, να ξαναφέρουμε κοντά μας αυτούς τους νέους που πρόωρα βρέθηκαν σε θέση επισφαλή. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των δασκάλων. Των δασκάλων ήδη στο δημοτικό, δηλαδή να ενισχύσουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα την κοινωνική παρακολούθηση. Είναι νέοι που έχουν γονεί σε επισφαλεί θέσει. Δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα παιδιά του. Στο σχολείο λοιπόν θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ένα παράγοντα κοινωνική ένταξη. Επιμένω πραγματικά εδώ στην κοινωνική αυτή παρακολούθηση, την κοινωνική συνοδεία κατά κάποιο τρόπο. Πρέπει να γίνει κατεπηγόντως κάτι ως προς αυτό. Έπειτα, για την απογοήτευση με τα πτυχία. Το είπε και ένας συνάδελφος και το επαναλαμβάνω και εγώ. Η απογοήτευση αυτή μας οδηγεί σήμερα στο να αναγκαστούμε να σκεφτούμε τον προσανατολισμό μας. Σήμερα πρέπει να πάψουμε να στέλνουμε τους νέους σε... σημεία, σε περιοχές όπου δεν θα προχωρήσουν. Τα πτυχία τους δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Πρέπει να μπορούν τα δικά τους σχέδια να τα προχωρήσουν, να τους ακούσουμε. Για τις νέες τεχνολογίες είναι πολλά αυτά που πολύ μεταβαλλόμενοι τομείς που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Η πράσινη τεχνολογία, οι νέες τεχνολογίες. Εκεί ως ε, Ευρωπαίοι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα ε, βοηθήσουμε ακριβώς να αναδυθούν αυτοί οι νέοι τομείς εργασίας. Έπειτα να κλείσω με δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, λέτε ότι είναι σημαντικό να λαφθούν υπόψη από κοινού η επαγγελματική πείρα και η εκπαίδευση. Ξέρετε εδώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν ταυτόχρονα να συγκεντρώνονται τις σπουδές τους και να δουλεύουν και στα McDonald's για να πετύχουν στη σταδιοδρομία του, Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε, εντάξει συμφωνώ με την επαγγελματική πείρα, δεν λέω, χρειάζονται να γίνονται τα στάζ όπω λέγονται, την περίοδο μαθητείας. Όμω θα πρέπει να είναι πολύ καλά πλαισιωμένα και αμοιβόμενα, διότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται τα στάζ ω πρόσχημα από τι επιχειρήσει, για να καλύψουν θέσεις εργασίας. Είναι μεταμφιεσμένες θέσεις εργασίας. Η δική μας ευθύνη λοιπόν ως βουλευτών και εκλεγμένων βουλευτών είναι οι νέοι να ανακτήσουν την αξιοπρέπεια, την αξιοπρέπειά τους, να πλαισιώσουμε ακριβώς αυτές τις περιόδους μαθητείας, τα στάζ και να ε, σταθώ στην ε, διακριτική μεταχείριση κατά την πρόσληψη. Όλοι οι νέοι που προέρχονται από περιβάλλοντα μειονεκτούντα ή από μετανάστες, επειδή έχουν ένα όνομα που ακούγεται ξένο, κατευθείαν είναι θύματα διακριτικής μεταχείρισης, με ή χωρίς πτυχίο. Ο δικός μας ο σκοπός είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες όλοι να έχουν ισότιμα δικαιώματα και όλες τις, ευ... τις ίδιες ευκαιρίες έναντι της αγοράς εργασίας. Δεν αρκεί να λέμε ότι να σεβαστούμε την οδηγία για μη διακριτική μεταχείριση. Εντάξει, συμφωνώ. Όμω πρέπει να επιβληθούν κυρώσει. Κυρώσει στι εταιρείε που δεν θέλουν να τι σεβαστούν τι οδηγίε. Πάρτε μια ε, συνοικία μειονεκτούσα, α πούμε, και αν η διεύθυνσή σα είναι εκεί, το όνομά σα ακούγεται ξένο, Υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Άρα όλοι αυτοί είναι ήδη εκτός κοινωνίας. λόγω καταγωγής, λόγω κατοικίας, περιοχής. Πού θα πάνε αυτοί οι νέοι. Θέλω πραγματικά λοιπόν να κάτσουμε και να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε ακριβώ αυτά τα θέματα. Να βρούμε πρακτικέ λύσει. Εγώ συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους, αλλά εδώ το σημείο αυτό είναι κατεπήγον, άκρος επίγον. Βλέπουμε μεγάλη απογοητεύση των νέων και ιδίω σε σχέση με όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ, πολιτικούς άνδρες και γυναίκες. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε κυρία Παπαδοπούλου. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ στα όσα έχει πει η κυρία ε, με την οποία είχαμε επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη και ειδικά των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Έχει Έχουν γίνει πολλές έρευνες και ακριβώς έχουν δείξει ότι τα επόμενα 10 με 20 χρόνια θα χρειαστεί ακριβώς επένδυση σε ειδικά προγράμματα για την νεολαία γιατί πραγματικά πρέπει να στηριχτούν οι νέοι, να έχουν κινητικότητα, να μπορούν τα επαγγελματικά επίπεδα κατάρτισης να αναγνωρίζονται από τη μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη και οπωσδήποτε να υπάρχει και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν για να καταπολεμηθεί η ανεργία ανάμεσα στους νέους. Όπως έχει τονιστεί σήμερα, οι νέοι μας διαθέτουν και πρώτον και δεύτερον και τρίτο πτυχίο. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν λιγοστέψει πολύ οι θέσει εργασία. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει στροφή ακριβώ προ τι πράσινε θέσει εργασία, για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, για θέσει που απαιτούν ψηλή τεχνολογική γνώση και καλή κατάρτιση και εδώ ακριβώ είναι που πρέπει να υπάρξει ένα ε, συντονισμό. Ε, σε λίγο χρονικό διάστημα, αρχέ του Δεκεμβρίου, θα δοθούν τα στοιχεία τη ΕΝΤΕΦΟΠ για να αποτελέσουν τη βάση για προγραμματισμό. Η δική μου η άποψη είναι ότι στα εθνικά στρατηγικά σχέδια θα πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα και προτεραιότητα στην νεανική επιχειρηματικότητα, πώ να βρεθούν πόροι για να μπορέσουν ακριβώ οι νέοι να αναπτύξουν εκεί που δεν μπορούν να μπουν στο δημόσιο να αναπτύξουν στον ιδιωτικό τομέα τι δικέ του επιχειρήσει. Η νεανική ε, η επένδυση στην νεανική είναι επιχειρηματικότητα νοσή σε αρκετέ χώρε, ιδίω στι νότιε χώρε, ενώ στις σκανδιναβικέ ή στην κεντρική Ευρώπη είναι σε καλύτερα επίπεδα. Και οπωσδήποτε ε, να καταπολεμηθούν οι διακρίσει. Θεωρώ ότι οι προκλήσει ε, που έχουμε ενώπιον μα είναι και προσκλήσει για να δούμε ακριβώ και τα εθνικά σχέδια πώς να αναβαθμίσουν τις προτεραιότητες τους για την νεολαία, για τις γυναίκες, για την κοινωνική ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών και από την άλλη χρειάζεται ένας συντονισμός ανάμεσα και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο σχολείο και στην οικογένεια. Ο συντονισμός πιστεύω ότι είναι η λύση σε πολλά προβλήματα. Thank you. Uh, before I ask uh, Mr. Martin to uh, Ευχαριστώ. Πριν ζητήσω από τον ε, κύριο Μάρκετ να απαντήσει να πω το εξή. Σε τι διαφάνειέ σα στην αρχή μιλήσατε για την ε, επισφαλή εργασία και λέτε ότι πολλοί δεν περνούν σε μια μόνιμη θέση επασχόλησης ε, στη συνέχεια. Υπήρξε μια έρευνα που έλεγε ότι οι περισσότεροι δεν το θέλουν. Το κατά πόσο ήθελαν να μείνουν άνεργοι σε επισφαλή εργασία Υπάρχουν και τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις, υπάρχουν ε, ε, και στη δική μου χώρα και σε άλλες χώρες που απογοητεύονται τόσο πολύ από όλο το σύστημα που τελικά αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να έχουν μία σταδιοδρομία στο μέλλον. Είναι πολύ διαφορετικά βέβαια τα πράγματα για πιο ειδικευμένου. Ήδη οι Γερμανοί συνάδελφοι ανέφεραν αυτό το θέμα. Άνθρωποι που μόλις βγήκαν από το πανεπιστήμιο και δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης για εκείνους. Επίσης, στην έρευνά σας έχετε διαπιστώσει κατά πόσο η επισφαλής εργασία μπορεί να είναι ένας τρόπος ε, να μπει κανεί σε μόνιμη εργασία. Γιατί έχω συζητήσει με συμπολίτε μου στην περιφέρειά μου γιατί και πολλοί μου έχουν πει ότι έχουν, έχουν, ε, θέλουν να, να, να κάνουν πολλές δουλειές πριν αποφασίσουν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα το λόγο σε εσά για 10 λεπτά το πολύ να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μοιραστούμε το χρόνο απαντήσεων ε, με τη συνάδελφό μου Σόνι θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά ζητήματα που επισημάνθηκαν πολλές φορές από όσους πήραν το λόγο. Καταρχάς το ερώτημα που ετέθη από την εισηγήτρια, που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είπε ότι αν οι κυβερνήσεις δώσουν κίνητρα στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν νέους, αυτό δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την ε, απασχόληση ε, στο σύνολό της. Όχι, αυτό είναι λάθος. Δεν υπάρχει πάλι μεταξύ των γενεών, μεταξύ των νέων εισαχθέντων στην αγορά εργασίας και των πιο έμπειρων εργαζομένων. Μόνο για το βραχύτερο χρονικό διάστημα υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και θα, το, θα τα δημοσιεύσουμε και στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης αλλά και στις επόμενες δημοσιεύσεις ε, που αφορά τις συντάξεις ε, με μια ματιά, αυτός θα είναι ο τίτλος, δεν υπάρχει μακροχρόνιος ανταγωνισμός μεταξύ νέων εργαζομένων και πιο έμπειρων εργαζομένων τα υψηλά ποσοστά, ε, οι χώρε που έχουν υψηλό ποσοστό απασχόληση έχουν και υψηλό ποσοστό νέων απασχολουμένων και το ίδιο ισχύει, αντίστροφα μάλλον, στι χώρε που δεν έχουν υψηλό ποσοστό απασχόληση. Λοιπόν, αυτό θέλω να το επαναλάβω γιατί είναι κάτι που το ακούω πολλέ φορέ ε, σε πολλές από τις διαδηλώσεις ε, στο Παρίσι σε σχέση με την μεταρρύθμιση για τις συντάξεις. Το δεύτερο που θα ήθελα να θέσω είναι το ερώτημα που μου ετέθη για τους κάτω του ελαχίστου μισθού, ε, μισθούς που έθεσε η συνάδελφος από την ε, Δανία. Καταλαβαίνω τους ενδιασμούς πολλών για το ζήτημα αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσει κανείς με τον εξής τρόπο. Ένα σύστημα μαθητείας καλά διαρθρωμένο, όπως αυτό που έχετε στη Δανία ή όπως αυτό που υπάρχει στη Γερμανία, στην Αυστρία, στις κάτω χώρες, ε, μερικές φορές, λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο όπως αυτό που προτείνω. Τον μισθό κάτω του ελαχίστου ξεκινάς ως ασκούμενος. Αν η αρχική σου παραγωγικότητα ε, είναι χαμηλή, έχεις και χαμηλότερη αμοιβή κάτω από τον ελάχιστο μισθό και όσο αυξάνει, ε, όσο περνάει ο καιρός και όσο αυξάνεται και η παραγωγικότητά σου, μπορεί ο μισθός σου να αυξάνεται επίσης. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτού και τη πραγματική σταδιοδρομία. Αν δούμε για παράδειγμα τι γίνεται στι κάτω χώρε, ξεκινά κανείς από την ηλικία των 15-16 ετών με έναν ελάχιστο μισθό που είναι το 30% ενός κανονικού μισθού και σιγά σιγά σύν το χρόνο αυξάνεται ο μισθός ε, ε, και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς για μένα αυτό είναι ένα καλά διαρθρωμένο σύστημα μαθητείας. Ε, εγώ σας λέω ποια είναι η δική μου άποψη, μπορείτε βέβαια να διαφωνήσετε. Τα στοιχεία που έχω ε, προέρχονται από τις χώρες που είναι πιο επιτυχείς ε, στα θέματα απασχόλησης. Κάτι ακόμη, συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε η κυρία Ντελή. Συμφωνώ απολύτως με το ότι σε σχέση με τις ομάδες που είναι οι πλέον ευάλωτες και στο πλαίσιο της κρίσης, αλλά και πέρα από αυτό, η ομάδα, οι ομάδες νέων που προέρχονται από λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον και που έχουν συσσωρεύσει πολλά μειονεκτήματα, το βασικό μας ε, η βασική μας αντιμετώπιση πρέπει να είναι έγκαιρη παρέμβαση. Και όταν λέω έγκαιρη εννοώ πριν πάνε στο σχολείο. Πρέπει να υπάρχει ισχυρή συνεχής επένδυση για την φροντίδα, την παιδική φροντίδα ε, για τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Υπάρχουν έρευνες που το αποδεικνύουν αυτό, ειδικότερα εάν η επένδυση συνεχιστεί ακόμη και αφού πάνε σχολείο. Και αυτό είναι το, το, το, σύστημα των συνοδευτικών μέτρων, ε, όχι μόνο δηλαδή για όλους όσους συμμετέχουν είναι εντός του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και για τις οικογένειές τους. Αυτό είναι μια σημαντική μακροπρόθεσμη ε, ε, επένδυση που πρέπει να γίνει και μάλιστα ακόμη και σε περίοδο κρίσης γιατί υπάρχει μια τάση περικοπών σε αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο της κρίσης. Τώρα, για την ομάδα των νέων που είναι η πλέον ευάλωτη είναι μια επένδυση η οποία θα έχει και τη μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό σας το λέω. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο να έχουμε αποτελεσματική παρέμβαση μετά που θα έχουν φύγει από το σχολείο, που θα έχουν παρατήσει το σχολείο οι άνθρωποι αυτοί. Τότε θα είναι πολύ αργά. Το τελευταίο θέμα που θα ήθελα να θέσω ε, σε σχέση με το συνδυασμό ε, δουλειάς και ε, σπουδών. Κοιτάξτε, θέσατε και το παράδειγμα του Αϊνστάιν. Πρέπει να σας πω ότι όταν δούλευε ήταν, ε, έκανε τις καλύτερες του ανακαλύψεις ο Αϊνστάιν. Αυτή ήταν η καλύτερη δουλειά του. Όταν παράλληλα ε, δούλευε και σε κάποια ε, δουλειά. Τότε ήταν η μεγαλύτερη παραγωγικότητά του. Και αυτό είναι κάτι που προκύπτει όχι μόνο από τις αγγλοσαξονικές χώρες, αλλά και από άλλες χώρες. Ο συνδυασμός δουλειάς και σπουδών, αυτή τη στιγμή βέβαια είναι μια δουλειά κάπως περιορισμένη, δεν μιλάω για πλήρη απασχόληση, δεν κάνει κανείς πλήρη απασχόληση τη στιγμή που, που σπουδάζει, γιατί αυτό είναι πραγματικά επιβλαβές για τις σπουδές, τους, για τις σπουδές του. Αν λοιπόν είναι πολύ σωστά διαρθρωμένη η διαδικασία, δουλειά και σπουδές, τότε βελτιώνεται και η ε, αποτελεσματικότητά τους μετά, όταν αρχίσουν τη σταδιοδρομία τους. Και τώρα θα ήθελα να σταματήσω εδώ και να δώσω το λόγο στη συνάδελφό μου για να απαντήσει σε ορισμένα από τα άλλα ερωτήματα που ετέθησαν. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια. Θα ήθελα να προβάλλω τα εξής σημεία. ΩΣΑ είναι ένα διεθνή οργανισμό. Συλλέγουμε αριθμητικά στοιχεία και πρακτικέ από πολλέ χώρε και δεν θα πούμε ότι η χώρα πρότυπο που όλοι πρέπει να παρακολουθήσουν η τάδε. Όχι. Περισσότερο θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε πρακτικές που υπόσχονται πολλά και είναι και καινοτόμε. Τέτοιε πρακτικές βοηθούν να επιληθούν προβλήματα όταν χρειάζεται κατεπηγόντω άμεσα και γι' αυτό έχουμε δώσει έμφαση στο χαρακτηριστικό της μάθησης. Διότι για όσους δεν, για τους νέους που δεν έχουν καλή σχέση με την εκπαίδευση, θέλουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για το μέλλον. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια θεωρητική, πειραματική προσέγγιση, πιλωτική, εκεί αξιολογούμε συγκεκριμένα μέτρα και προσπαθούμε να προωθήσουμε κάποια βασικά μηνύματα. Μηνύματα τα οποία δεν πρέπει να υλοποιούνται αυτομάτως από τις χώρες, πρέπει να λαμβάνουν θέση οι χώρες έναντι των μηνυμάτων αυτών. Έχουμε λοιπόν ειδικέ συστάσεις χώρα, όπως συχνά συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν πάρουμε λόγου χάρη την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αυτή του είδους εκπαίδευση έχει πολύ ε, μεγάλη αξία για χώρες και τους δίνουν ιδιαίτερη έμφαση. Οι γονείς και τα παιδιά κάνουν πολλά για τους γονείς, για τα, οι γονείς κάνουν πολλά για τα παιδιά τους μάλλον, αλλά όχι προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την ε, εικόνα που έχει η επαγγελματική εκπαίδευση στη Γαλλία. Πρόσφατα έπρεξε μια μεγάλη επανάσταση. Ε, ένας ένα μεγάλο λεωφορείο, μια βασιλική οδό θα έλεγα από τους, ε, στα σχολεία για να κατευθυνθούν οι μαθητές προς αυτήν την ε, επιλογή για να χρηματοδοτούν τις σπουδέ τους, να δουλεύουν σε εργαστήρια ως μαθητευόμενοι αλλά να γίνουν ε, και μηχανικοί αν έχουν ιδιαίτερα προσόντα, είναι ταλαντούχοι και ούτω καθεξής. Μπορούμε λοιπόν να μεταφέρουμε πρακτικές από μια χώρα στην άλλη. Με τρόπο σχετικά απλό. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Έπειτα, ο δυναμικό χαρακτήρα είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό μου άρεσε πολύ το σύνθημά σα, το μήνυμά σα τέλο πάντων. Η νεολαία εν Γιατί θα πρέπει οι νέοι να μην ε, βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα τέλμα, ούτε να φυλακίζονται από επισφαλίστε εργασία. Πρέπει να φροντίσουμε να μην είναι μόνο τους επιλογή η μερική απασχόληση. Βλέπουμε σε κάποιες χώρες ότι ναι, ξεκινούν από επισφαλείς θέσεις, αλλά αυτό τουλάχιστον είναι καλύτερο από το να ξεκινήσει κανείς από την ανεργία. Γιατί έτσι ανοίγουν οι πόρτες για κάποιους νέους, για αρκετούς νέους. Συχνά δράση πρέπει να αναλυφθεί προηγουμένως Γι' αυτό λοιπόν η απασχόληση πρέπει να συνδυαστεί με την εκπαίδευση ήδη από τα φοιτητικά χρόνια των νέων. Πρέπει η παρακολούθηση να γίνει από τη στιγμή τη ε, φοιτητική σταδιοδρομία. Πριν περάσει κανεί στην αγορά εργασία. Πριν έρθει αντιμέτωπο με αυτή την αγορά. Τελευταία παρατήρηση, και αυτό είναι ένα στοιχείο που ε, το προβάλαμε ιδιαίτερω στο φόρουμ του Όσλο. Η συμμετοχή όλων των παραγόντων είναι σημαντική, ιδίω σε τοπικό επίπεδο. Εάν κοιτάξετε τον ιστοτοπό μας είχαμε παρουσιάσεις από παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην ε, πράξη και μας είπαν τι μπορούν να κάνουν εκείνοι, τι κάνουν εκείνοι οι ίδιοι για τους νέους. Γι' αυτό και το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό για να κινητοποιήσει όλους τους τοπικούς παράγοντες, πράγμα που έγινε στα, στις σχολές δεύτερη ευκαιρία, όπω λέγονται, όπω αυτό που επισκεφτήκαμε στη Μασαλία και λειτουργεί με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα πρέπει όλοι να αισθανθούν αυτήν την ε, ανάγκη. Οι νέοι ίδιοι συμπεριλαμβανόμενοι. Οι εργοδότες μπορούν να κάνουν κάτι για τους νέους, ακόμα και σε αυτή την περίοδο κρίσης. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Ευχαριστούμε κύριε Μάρτιν. Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σα. Ήταν πολύ χρήσιμη συζήτηση. Ξέρω ότι άρεσε και στου συναδέλφου. Σα ευχαριστώ ξανά. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, έκθεση 2010 για την υλοποίηση των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2007-2013. Να δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω στα αγγλικά. Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να συστήσουμε στην Επιτροπή, να προτείνουμε την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ως ε, υπεύθυνη επιτροπή για να υλοποιήσει τι συστάσει από την Επιτροπή Απασχόληση Κοινωνικών Υποθέσεων σε αυτό το σχέδιο ψηφίσματο. Πρώτα απ' όλα, καλωσορίζουμε την στρατηγική έκθεση τη Επιτροπή για την υλοποίηση τη πολιτική συνοχή και των σχετικών προγραμμάτων, όπω συγχρηματοδοτούνται από το Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2007-2013. Υπογραμμίζουμε ότι αυτή η στρατηγική έκθεση είναι ένα νέο στοιχείο τη πολιτική συνοχή, το οποίο εισήχθη από τον κανονισμό του Συμβουλίου το 2006. Ε, καλωσορίζουμε το γεγονό ότι αυτή η επισκόπηση αντιμετώπιση βασίζεται στις εθνικές στατικικές εκθέσεις 27 κρατομελών επειδή με την διαδικασία αυτή έχουμε βελτιώσει αισθητά την διαφάνεια και το υπόλογο, τη λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, ε, ελέγχουμε την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του κάθε κράτου μέλου και το τι πρόοδο έχει επιτελεστεί σε εθνικό επίπεδο ό,τι αφορά την υλοποίηση των στατικικών κατευθυντηρίων γραμμών. Θεωρούμε ωστόσο ότι με μετά την διεθνή οικονομική ύφεση, η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να παρέχει μια ενδελεχέστερη παρουσίαση του αντικτύπου των τομέων που καταμετρήθηκε η πρόοδο. Δηλαδή, ω προ την δημιουργία νέων θέσεων εργασίων, εργασία, την κάλυψη των οικονομικών κοινωνικων διαφορών, την ανεργία και άλλα στοιχεία. Αυτό είναι καθοριστική σημασία γιατί κατά την άποψή μα το οικονομικό σκηνικό, οικονομικό τοπίο έχει αλλάξει δραματικά μετά την οικονομική κρίση του 2008. Η οικονομική αύξηση έχει ε, περιοριστεί, η απασχόληση συρρυκνώθηκε, ε, οι επενδύσεις μειώθηκαν και υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Ε, υπάρχουν λοιπόν νέες ανάγκες που παρουσιάστηκαν, νέες προτεραιότητες, όλα αυτά λοιπόν απαιτούν οι χώρες ε, στα στρατηγικά εθνικά τους προγράμματα να ε, λάβουν υποψηφιά αυτά στοιχεία και τους εθνικούς κοινοτικούς στόχους για καλύτερες ε, θέσεις εργασίας, την κοινωνική ανάκαμψη, την ενσωμάτωση, την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινοτομία. Οι υπόλοιπε συστάσεις μας είναι ότι καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει ήδη γίνει στην υλοποίηση προγραμμάτων για τι περισσότερε και καλύτερε δουλειέ, τη σχετική κατευθυντήρια γραμμή δηλαδή, και συστήνουμε εντόνω η κινητοποίηση των ε, κονδυλίων για την επίτευξη των στόχων καταπολέμηση τη ένδυα στα πλαίσια του στρατηγική τη Ευρώπη του 2020 θα πρέπει να γίνει ένα στόχο προτεραιότητα. Επισημαίνουμε ότι ακόμη Και αν καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει επιτελεστεί, σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να έχουμε ε, ε, λεπτομεριακά δεδομένα για τον αντίκτυπο που υπήρξε ω τώρα, διότι αυτά θα είναι διαθέσιμα μόλι το 2012. Επίση, καλούμε τα κρατημέλη να μειώσουν την το υπέρμετρο διοικητικό κόστο και του φραγμού που εμποδίζουν την επίτευξη πολιτικών στόχων για την πρόσβαση στην ε, απασχόληση, την καταπολέμηση τη ένδυα και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων. Θεωρούμε ότι το, η πειθαρχία και η στοχοθεσία βελτίωσε την υλοποίηση των προγραμμάτων. Η βιώσιμη και η συμμετοχική ανάπτυξη είναι μια από τι προτεραιότητε τη Στρατηγική τη Ευρώπη του 2020. Κατά συνέπεια, όλα τα έθνη, όλα τα κρατημέλη πρέπει να αποφύγουν τι καθυστερήσει στην επιλογή και την υλοποίηση προγραμμάτων στο μέλλον. Θα πρέπει να μειώσουν και την γραφειοκρατία και υπάρχει σαφής ανάγκη να προαχθεί μια πιο πράσινη, πιο ανταγωνιστική και πιο αποτελεσματική ως προς την κατανάλωση των πόρων πολιτική. Η κοινωνική και η συνοχή να προαχθεί σοβαρά. Επίσης καλούμε στην γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή να προωθήσει την αποτελεσματικότητα του ε, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με τα κονδύλια του ώστε να επιτευθούν στόχοι που θα επιτρέψουν στους Ευρωπαίους πολίτες να γίνουν απασχολήσιμοι και προσαρμόσιμοι δεδομένων των συνθήκων που έχουμε θέσει και των όρων που έχουμε θέσει για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο προκειμένου να προαχθεί η Ευρωπαϊκή Στατική του 2020 για τις θέσεις εργασίας και την απασχόληση. Ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία λοιπόν στον τρόπο που το Ταμείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ώστε να καλυφθούν οι διαφορές στην ευημερία και τις συνθήκες διαβίωσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης για να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες των πολιτών και να έχουν καλύτερες προοπτικές στις θέσεις εργασίας. Πιστεύουμε ότι αυτό το Ταμείο, το κοινωνικό, είναι ένα εργαλείο για να καταπολεμηθεί είναι ο κοινωνικό αποκλεισμό και η ανεργία και γι' αυτό καλούμε την Επιτροπή να ενισχύσει το δυναμικό του ΕΚΤ, την οικονομική του αυτονομία και την ευελιξία του, προκειμένου να πλουστευτούν οι διαδικασίε, η παρακολούθηση και η έλεγχη. Θα πρέπει Τέλος, η Επιτροπή να ενισχύσει την παρακολούθηση της προοδού και την καταμέτρησή της επιβάλλοντας την ε, χρήση βασικών δικτών στι στις εθνικές εκθέσεις τις στρατηγικές εκθέσεις. Θα πρέπει να υπάρχει σύγκληση όλων των πολιτικών στόχων και των αποτελεσμάτων τους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τις ε, κοινωνικές ευκαιρίες και την στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Η χρήση των βασικών δικτών μπορεί να βελτιώσει την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου σε εθνικό επίπεδο. Καταλαβαίνω ότι η γνωμοδότηση αυτή ε, επιδέχεται τροπολογιών με μια προθεσμία που νομίζω έχει οριστεί στις 15 Νοεμβρίου. περιμένουμε εναγωνίως τις τροπολογίες σας, διότι έχουμε χρονικούς περιορισμούς και ε, περιορισμούς προς τους χαρακτήρες, 200 χαρακτήρες για την έκθεση, οπότε θέλουμε να δούμε και τις τροπολογίες σας για να δούμε πόσο, η έκταση θα καλύπτει η έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κυρία Φιγκερέιδο. Κυρία Σέτρο πρώτα. Για τελευταία φράση της συγκήτριας ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα τη βοηθήσουμε ώστε να έχουμε ως το δυνατόν ευρύτερη γρομοδότηση. Σας δεν βεβαιώ γι' αυτό. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε πού υπάρχει αυτό το κείμενο της Επιτροπής, ποιες είναι οι θέσεις του, γιατί έρχεται με τόση καθυστέρηση. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με την επαλήθευση των λειτουργικών προγραμμάτων που είναι καλή, αλλά με το έγγραφο πλαίσιο, το εθνικό έγγραφο πλαίσιο για τα ερωτικά ταμεία που ουσιαστικά θα έπρεπε να έχει κατευθεί το 2008 και έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση. Και η Επιτροπή χρειάστηκε ώρε για να μα το ετοιμάσει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν καλό για άλλη μια φορά να διατυπώσουμε τι επικρίσει μα και να επιμένουμε. Διότι τελικά το έγγραφο αυτό δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα πλέον. Εν τω μεταξύ έχει αλλάξει η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Αύριο θα έχουμε και την έκθεση συνοχής ε, που θα μας υποχρεώσει να κοιτάξουμε παραπέρα και έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον πιστεύω να δούμε πώς έχουμε φτάσει, ε, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε από το χαμηλότερο επίπεδο και πέρα. Επίσης θα πρέπει να δούμε αν ήταν καλά τα αποτελέσματα ή όχι και αν τα κράτη-μέλη αξιοποίησαν τα προγράμματα αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπετε πώ τώρα μέσα προβλέπονται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, πρόγραμμα δεν έχουν ε, αξιοποιηθεί ικανοποιητικά από τα κράτη-μέλη. Είναι μάλλον περιορισμένη η αξιοποίηση που διαπιστώνεται. Και εγώ τουλάχιστον από τη Γερμανία είμαι σε θέση να γνωρίσω ότι πολλά από τις, πολλές από τις ευκαιρίες, που υπήρχαν δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό και να αναφέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένα πράγμα είναι το gender budgeting, ιδιαίτερη έμφαση στο φύλλο μέσα, ε, στην διάσταση του φύλου μέσα από τον προπολογισμό. Αυτό δεν το επαλήθευσε καν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μια φράση που λέει ναι, στρατηγική πλαίσιο θα μπορέσει να περάσει μέσα από τα λειτουργικά προγράμματα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το καθήκον να μεριμνήσει για το gender budgeting. Αυτό ήταν όλο. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέραν αυτή τη φράση στο έγγραφο και μου φαίνεται ότι είναι σκάνδαλο κάτι τέτοιο. Έχουμε αγωνιστεί για μια τέτοια παράγραφο και θα θέλαμε κάτι περισσότερο. Δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε μια απλή αναφορά. Θετικά, Τώρα συμβιώνω ότι ε, το άρθρο 5 φαίνεται να φέρνει καρπού. καρπούς. Πρέπει να το πούμε και στην Επιτροπή. Αλλά γιατί άλλα μέσα όπως ε, την ε, συνολική επιδότηση δεν τα αξιοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε καλά παραδείγματα που θα μπορούσαν να έχουν βοηθήσει. Υπάρχει μια σημαντική παράγραφος η οποία λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προαγάγουν ε, εφάνταστα ή δημιουργικά προγράμματα και διεθνικά προγράμματα που όμως δεν υλοποιήθηκε και σε αυτό δεν κάνει κανένα σχόλιο η επιτροπή. Και ένα άλλο σημαντικό σημείο το οποίο βλέπουμε όσο ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά καθημερινά είναι ότι υπάρχουν χαμηλές προκαταβολέ από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι απαγορευτικέ για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, εκείνε οι οποίε δεν είναι σε θέση καν να καταθέσουν πρόταση, γιατί δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσουν την έλλειψη σε χρήματα που δεν του έχουν προσφερθεί, δεν του έχουν προκαταβληθεί. Δεν είναι σε θέση δηλαδή να μείνουν χωρί πληρωμέ αυτέ οι μη κυβερνητικέ οργανώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δεν μπορούν καν να επιβιώσουν τελικά αυτέ οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, ναι, ίσω να μην είναι ε, γενικευμένο, αλλά πάντω έχει μεγάλη σημασία. Το earmarking επίσης βλέπουμε ότι λειτουργεί ικανοποιητικά. Βλέπουμε ότι έχει επιδείξει μεγάλη ευελιξία το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε σχέση με την ε, κρίση. Και μπορώ να πω ότι ναι, καλή ευελιξία, αλλά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση δεν χρειαζόμαστε earmarking, χρειαζόμαστε σαφείς δείκτες, σαφείς ε, σαφείς μονάδες μέτρησης, τις οποίες άλλωστε ανέφερε η συγκήτρια και με πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Φιγκερέιδο. Κυρία Φιγκερέιδο. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Ιδίως το πώς ε, αξιοποιούνται τα κονδύλια και σε σχέση με την ίδια την πολιτική της συνοχής και τα υπάρχοντα προγράμματα. Να θυμίσω εδώ ότι πέραν κάποιων παρατηρήσεων που ήδη διατυπώθηκαν, να θυμίσω λοιπόν ότι υπήρχαν προγράμματα, ιδίως στον τομέα της ισότητας των δικαιωμάτων, όπως το Equal, που όταν ολοκληρώθηκαν ε, προκάλεσαν σχόλια όπως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο θα συμπλήρωνε τα αποτελέσματα. Για την ώρα δεν έχουμε αυτές τις απαντήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, τα συμπληρώματα. Υπάρχουν πολλοί τομείς που από αυτή την σκοπιά σχετίζονται με το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα άλλα διαρθωτικά όπω το ίδιο το Ταμείο Συνοχή, με το πώς λοιπόν χρησιμοποιούνται. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ακριβώς και η διάσταση της ισότητας των ευκαιριών, των δικαιωμάτων μάλλον. Ιδίω από την άποψη των φίλων της ισότητας των φίλων Ήθελα πάντως να πω ότι ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολλές χώρες, ιδίως Όσε έχουν πιο αδύναμες οικονομίες και δημοσιονομικές καταστάσεις ευάλωτε, και όπου η διοργάνωση των χωρών αυτών των ίδιων δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε εθνικό επίπεδο επαρκώς σε κοινού στόχου για να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα διαφορετικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχή. Αυτοί λοιπόν που έχουν τι περισσότερε ανάγκε και τη μεγαλύτερη αδυναμία έχουν και τι περισσότερε δυσκολίε. Αυτό επιδεινώνει την ε, ύπαρξη διαφορών. Και καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή, εκταμιεύουμε κονδύλια από τα ταμεία αυτά βάσει των κανόνων τους και κατευθύνονται σε οργανώσεις και θεσμικά όργανα, αλλά σε χώρες που με προπολογισμό, με τον προϋπολογισμό που διαθέτουν, δεν μπορούν να συμπληρώσουν τα κονδύλια αυτά ώστε να χρησιμοποιηθούν αρκετά. Οπότε υπάρχει μια μετατόπιση των κονδυλίων και επιδεινώνονται οι διαφορές. Ε, το αποδεικνύει η ίδια πραγματικότητα ότι αυτά συμβαίνουν. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να ακούσω και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εκτίμησή της. Όπως υπόθηκε εδώ, θα θέλαμε να υπάρχει προσεκτικότερη ανάλυση όλων αυτών των θεμάτων. Περισσότερα από όσα έχουμε ήδη επιτάπτους. Διότι η εξέλιξη των πραγμάτων δυστυχώς και γρήγορη είναι και αρνητική κατεύθυνση έχει. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε κατεπηγόντως, με κατεπήγοντα καθαρακτήρα τις επιταγές των ταινίων. Νομίζω λοιπόν ότι κάποιε από αυτέ τι επισημάνσεις καλό είναι να αναφέρονται και στην ίδια μα την αναδότηση. Ε, Το είπε και η συγκεκριά μα. Ήδη έχουν γίνει πολλέ ε, σωστέ κινήσει Με τι τροπολογίε μα ελπίζουμε να συνεισφέρουμε επαρκώ, να συμπληρώσουμε τη λύπη και να προτείνουμε και πρόσφορε λύσει. ώστε η έκθεση να λάβει τη μορφή που θέλουμε και να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Ε, είναι κατεπίγοντα τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιασλοβιέσκα και μετά η κυρία Γκρινή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ως γενική παρατήρηση θα ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Ζητείται ευελιξία και καλύτερο έλεγχος ε, των ε, εξόδων και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Όμως υπάρχουν κάποιες ανεπάρκειες όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, κατά την άποψή μου. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Απασχόληση δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει με τον να κάτι τέτοιο από την εκνομοδότηση αυτή. Ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι η αξιολόγηση της ε, αγοράς εργασίας. Η σχέση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και των ε, μακροοικονομικών συνεπειών είναι δύσκολο να καταδειχθεί, γιατί είναι δύσκολο να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτό που πραγματικά θα έχει επίδραση είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και αυτό είναι δύσκολο να το μετρήσει κανείς. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να ε, δοθεί έμφαση στα μέτρα καταπολέμησης της κρίσης. Τώρα, η καταπολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα σύμφωνα με τη γνωμοδότηση. Κοιτάξτε, εγώ ε, δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι το ε, ταμείο αυτό πρέπει να επιτύχει, να προσπαθήσει να επιτύχει τους στόχους Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και όχι να επιμείνει μόνο στην καταπολέμηση της φτώχειας. Αν προσπαθήσουμε πάρα πολύ να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, ενδεχομένως ε, μπορεί να καταλήξουμε τελικά στο αντίθετο αποτέλεσμα. Καλύτερα θα ήταν ε, να ε, συμμετέχει περισσότερο η κοινωνία του πολίτη, να ε, προάγουμε το επιχειρήν. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Ιδιαίτερα τονίζεται επίσης ο ρόλος της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Νομίζω ότι το Ταμείο αυτό θα έπρεπε να αξιολογεί ε, περισσότερο την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης και το λέω αυτό σε σχέση με την εμπειρία που έχουμε ε, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής όσον αφορά τώρα την ε, οικονομική ανεξαρτησία, την αυτονομία του συγκεκριμένου ταμείου, νομίζω ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω με, το να θεωρηθεί κάτι ξεχωριστό αυτό το ταμείο από την πολιτική συνοχή. Η πολιτική συνοχή πρέπει να εφαρμόζεται σε ένα σύνολο δράσεων. Μιλήσαμε ήδη για τη συμπληρωματικότητα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όσον αφορά το σημείο 6, προτείνεται μια αλλαγή νοοτροπίας να μην έχουμε μόνο input, να έχουμε και outcome και συμφωνώ απολύτω. Η κυρία Γκρινή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ω εισηγήτρια για το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προφανώ έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για αυτό το κείμενο. Δεν είχα ακόμα τον καιρό να το μελετήσω εντελεχώ. Θα φροντίσω όμω να υποβάλω τροπολογίε και όπω και η προηγούμενη συνάδελφο, Πιστεύω ότι πραγματικά εδώ υπάρχει μια διασύνδεση με την καταπολέμηση της φτώχειας και με πολλά άλλα στοιχεία που επηρεάζουν και τη στρατηγική του 2020. Δεν θα πρέπει όμως το κείμενο να μετατραπεί σε κείμενο για την καταπολέμηση της φτώχειας. Εγώ παρόλα αυτά έχω το εξή μήνυμα. Ναι στην καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά με κοινωνική ένταξη. Δηλαδή απασχόληση. Αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως. Ε, προσοχή λοιπόν για τους στόχους και των προγραμμάτων αυτών για την ποιότητα της εργασίας. Ε, υπάρχουν πολλά στοιχεία εδώ που πρέπει να τα προσέξουμε. Θα φροντίσω λοιπόν να αποστείλω στην συνάδελφο τις τροπολογίες μου. Την ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή που θα τους δώσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται κανείς να ζητά το λόγο, οπότε το λόγο έχει πάρει η κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ όλες τις αδέρφους που έχουν πάρει τον λόγο. Θεωρώ ότι τέθηκαν επιτάπητος πολύ σημαντικά θέματα. Θα συμφωνήσω με την κυρία Σρότερ που έχει πει ότι το έγγραφο δεν κατατέθηκε έγκαιρα. Είναι γεγονός ότι καθυστέρησε το έγγραφο και αυτό μπορεί να το υποδείξουμε στην Επιτροπή. Ε, σίγουρα έχετε επισημάνει ότι η κατάσταση έχει αλλάξει από το 2008. Είναι αυτό που, που και εγώ έχω αναφέρει. Πολλά έχουν αλλάξει από το 2008 μέχρι το 2010 και διαφορετικά τα βιώνουν οι πολίτες σε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συμφωνώ ότι κάποια κράτη έχουν αξιοποιήσει κάποια προγράμματα και κάποια άλλα όχι. Ε, ακριβώς εδώ είναι που πρέπει να επικεντρωθούμε ώστε όταν καταρτίζονται τα εθνικά στρατηγικά προγράμματα να υπάρχουν συγκεκριμένες προτεραιότητες που να συνάδουν ακριβώς με όλους τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Και εδώ απαντώ και στις δύο τελευταίες συναδέλφους. Ε, αν εδόθηκε περισσότερη βαρύτητα στη φτώχεια είναι γιατί ακριβώ διανύουμε φέτο και το έτο 2010 που είναι για την καταπολέμηση τη φτώχεια. Δόθηκε ειδική έμφαση σε αυτόν τον στόχο, Αυτό όμω δεν αποκλεί και όλου του άλλου στόχου τη στρατηγική 2020 που αφορούν και καλύτερε θέσει εργασία και περισσότερη εμπλοκή των γυναικών και αυτό μπορεί μέσα από τα amendments μα, τι τροπολογίε μα, να μπει στην έκθεση. Όπω έχω πει, όταν ε, πρέπει να περιοριστεί σε 200 χαρακτήρες δεν μπορείς να ενσωματώσεις όλες τις απόψεις. Για τον gender budgeting συμφωνώ και υπερθεματίζω, γιατί θεωρώ προσωπικά ότι ήταν μια πρωτοβουλία της Γερμανικής Προεδρίας και σίγουρα θα έπρεπε να ενισχυθεί και στις επόμενες Προεδρίες. Κάτι που εγώ προσωπικά βλέπω ότι δεν έχει γίνει. Το gender budgeting είναι ο μόνος πρακτικός τρόπος κατά την άποψή μου που μπορεί ακριβώς να πιέσει τις κυβερνήσεις όταν καταρτίζουν εθνικούς προϋπολογισμούς να εντάξουν όχι μόνο προγράμματα και λεφτά για να χρηματοδοτήσουν ε, projects για τη γυναίκα και την ισότητα, αλλά να κάνουν monitoring της, προ... πρόοδου. Να κοιτάζουν τι ακριβώς αποτελεσματικότητα έχουν τα συγκεκριμένα λεφτά μέσα στους προϋπολογισμούς για να φέρουν αποτελέσματα. Ε, όσον αφορά το... για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχει λεχθεί ότι παίρνουν χαμηλέ προκαταβολέ. Αυτό είναι γεγονό. Και αυτό να αποκλεί μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, από το να επιβιώσουν και να ασκούν τον ρόλο που πρέπει. Και αυτή είναι μια πολύ σωστή επισήμανση. Για του δείχτε, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, όλοι συμφωνούμε ότι σωστά ζητούμε να μπουν σαφεί δείχτε και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Όσον αφορά δε το Ευρωπαϊκό ε, Κοινωνικό Ταμείο, όπω έχει πει η κυρία Φικερέιδο, ε, ναι, αναμέναμε ότι θα συμπληρώσει κενά τα οποία δεν καλύφθηκαν από προγράμματα όπως το Equal. Το Equal. Αυτό δεν έχει γίνει και πιστεύω ότι μπορεί μέσα από τις τροπολογίες να πούμε ακριβώς ότι πρέπει να χρηματοδοτεί όσους έχουν περισσότερη ανάγκη και ανάμεσα σε αυτούς που έχουν ανάγκη είναι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται ανάμεσα σε άλλα και σε θέματα της ισότητας των φύλων. Τέλος, ε, η αναφορά που έγινε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πω και εγώ ότι συμφωνώ ότι πρέπει να είναι πιο ευέλικτο, να γίνεται καλύτερο έλεγχο των εξόδων, να αξιολογείται η ποιότητα των θέσεων εργασία και εδώ ακριβώ θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα ε, και στο σωστό επιχειρήν και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να αξιολογηθεί ώστε όλε οι όλοι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 να μπορέσει μέσα από τα προγράμματα και τα εθνικά στρατηγικά σχέδια να υλοποιηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 15 Νοεμβρίου το μεσημέρι και η έγκριση στην Επιτροπή θα είναι στις 2 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για όλα αυτά κλείνουμε με τη συνεδρία τη Επιτροπή για σήμερα. Σα ευχαριστώ. Ω, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια ειδική συνάντηση στο Στρασβούργο. Έκτακτη. Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, 7 με 8.30. Συνάντηση και στο Στρασβούργο τη Δευτέρα.